Αγαπητοί συνάδελφοι, σας προτείνω να ξαναρχίσουμε και μάλιστα να μην καθυστερήσουμε καθόλου γιατί έχουμε πολύ βεβαρημένη ημερήσια διάταξη. Πολλά πράγματα έχουμε. Θα δώσω τον λόγο στη Γιούτα Στάινροπε για να μας δώσει ε, μία, έτσι, ε, ε, να μας πει τι γίνεται με τον τριμερή διάλογο ψή. Από ό,τι φαίνεται δεν θα, έχει, δεν θα αλλάξει ο τίτλος. Να μας πει λοιπόν τι συμβαίνει εκεί. Είναι το μόνο σημείο το οποίο ήταν εγγεγραμμένο ήδη στη μέρη διάταξη της πρωινής, ε, ε, συγγνώμη ήταν εγγεγραμμένο το πρωί και δεν καταφέραμε να το α, συζητήσουμε. Σας είπαμε ότι επανειλημμένα ζητήσαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναφερθεί σε μια πρωτοβουλία η οποία έχει ξεκινήσει έτσι ώστε να επικαιροποιηθεί ε, το Γιούρες στα πλαίσια του ΨΥ. Ε, το κείμενο από ό,τι φαίνεται έφτασε χτες και εξεκολουθεί να υπάρχει πρόβλημα. Γι' αυτό λοιπόν Θα δούμε. Θα έχουμε αύριο μια επαφή ξανά, θα έχω εγώ με την Επιτρόπο για να δούμε πώς μπορούμε να, με τον Επιτρόπο μάλλον, για να δούμε ε, πώς μπορούμε να συνεχίσουμε τα πράγματα και τη διαδικασία και βεβαίως όλα αυτά ε, θα σας ε, αναφερθούν εν λεπτομερία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Καταρχάς να ευχαριστήσω όλους όσους συμμετείχαν ε, από το Κοινοβούλιο στον τριμερή αυτό διάλογο. Είναι, ήταν πολύ σημαντικό να εργαζόμαστε όλοι προς την ε, ίδια κατεύθυνση, έτσι ώστε να μπορέσουμε να βρούμε μαζί συμβιβασμού, τους οποίους θα ψηφίσουμε σε αυτήν την Επιτροπή και θα προσπαθήσουμε να τους μεταφέρουμε. Αυτό το είδα και από την ε, ιδιότητά μου ως κοιόδηση ή Από την πλευρά του Συμβουλίου την περασμένη Πέμπτη συζητήσαμε το κεφάλαιο μικροχρηματοδότηση κοινωνική ε, κοινωνικές επιχειρήσεις. Ήταν θετικά τα αποτελέσματα για εμάς, για το Κοινοβούλιο. Είχαμε 45% συμμετοχή μικροχρηματοδότηση και κοινωνική, ε, κοινωνικές ε, επιχειρήσεις. Έχουμε δώσει βάση στους, ε, σε αυτούς που βρίσκονται σε μειονεκτική κοινωνικά θέση και προσπαθούμε να διασφαλίσουμε, για παράδειγμα, κατάρτιση και απόκτηση δεξιοτήτων μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Συζητήσαμε για τις πράξεις κατά εξουσιοδότηση, ε, το οποίο είναι ένα θέμα προτεραιότητας, ε, είναι μια οριζόντια, ένα οριζόντιο θέμα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και στο σύνολο των διαπραγματεύσεων πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντική για μας η θέση του Συμβουλίου. Η θέση του Συμβουλίου είναι κάτι που δεν μπορούμε να δεχτούμε και περιμένουμε περαιτέρω συζητήσει. Επίση, την περασμένη εβδομάδα αρχίσαμε να ζητούμε το κεφάλαιο Γιούρε και για μένα είναι λυπηρό ότι το Συμβούλιο έχει τέτοια θέση. Ήταν πολύ... Θα ήταν πολύ πιο εύκολο να συζητήσουμε εάν μπορούσαμε να ανταλλάξουμε επιχειρήματα με ε, και με την συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι κάπως ακλόνητη και έτσι εμείς ε, με το ρόλο του νομοθέτη το Συμβούλιο και με το Συμβούλιο πρέπει να βρούμε μια συμβιβαστική λύση σίγουρα. Ένα σημαντικό σημείο για εμάς είναι το ποσοστό συμμετοχής ε, στις συνοριακές συνεργασίες. Εδώ όμως δεν υπήρξε κάποια συμφωνία, δυστυχώς. Την Δευτέρα παρουσιάστηκε η μεταρρύθμιση της Γιούρες. Υπάρχουν ε, αλληλοεπικαλύψεις, ιδιαίτερα για το θέμα της Γιούρες, τη Άξο και ως ε, εισηγήτρια να πω ότι είμαι έκπληκτη με τα αποτελέσματα αυτά των διαπραγματεύσεων. Ένα σημείο θα ήθελα να αναφέρω διότι με έχει εξοργήσει. Εάν όλοι εμείς οι εισηγητές στην Επιτροπή Απασχόλησης θέλουμε να έχουμε μια κοινή θέση έξω από αυτό το κοινοβούλιο. Ε, θα, να σας πω ότι η εικόνα που δίνουμε είναι ότι το κοινοβούλιο δεν ξέρει πού βρίσκεται, ότι δεν έχει κάποια ενιαία θέση. Και τη χρειαζόμαστε αυτή, διότι έτσι θα πετύχουμε και ε, περισσότερο σεβασμό Στις 6 Νοεμβρίου διεξήχθηκαν συζητήσει ε, με την Συντονιστική Επιτροπή για το Γιούρες και πιστεύω πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενδιαφέρθηκε να μάθει τι έγινε ε, στις συζητήσεις εδώ στο Κοινοβούλιο και όσον αφορά τις ε, συνοριακές ε, συνεργασίες, πιστεύω ότι αυτό μας φέρνει πιο κοντά σε ένα αποτέλεσμα. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να κάνουμε σχόλια. Ακούσαμε, είχαμε αυτήν την πιστή αναμετάδοση όλων των στοιχείων. Νομίζω ότι θα πράξουμε τα δέοντα. έτσι ώστε και το σύνολο του Κοινοβουλίου ε, να γνωρίζει βέβαια και τι γίνεται με τις διαπραγματεύσεις που όπως λέει και η συγγήτρια ε, παραμένουν πιστές στην εντολή που έχουμε δώσει εμείς και το σύνολο των πολιτικών ομάδων. Ωραία, τελειώσαμε με αυτό το σημείο. Ε, τώρα φτάνουμε στο σημείο 10. Το σημείο 10 λοιπόν, βάσει του οποίου θα πρέπει να συζητήσουμε την έκθεση της συναδέλφου Ντανούτα Γιασλόφκιακα σχετικά με την οδηγία που αφορά την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παραχής υπηρεσιών. Θα δώσουμε το λόγο λοιπόν στην κυρία Γιασλοβίτσκα για να παρουσιάσει την έκθεσή της. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ ε, κυρία Πρόεδρε. Μετά από 16 χρόνια από την, ε, την ε, έγκριση της οδηγίας 9671 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας παρουσίασε μια οδηγία που αφορά την επιβολή της οδηγίας 9671. Λοιπόν, πρόεδρος ε, διακόπτει την, ε, ε, την ομιλήτρια και λέει ότι να μιλάτε με έναν αριθμό κανονικό έτσι ώστε να μπορούν να σας ακολουθήσουν και οι διερμηνείς. Πάρα πολύ ωραία. Ναι, ζητώ συγγνώμη. Ζητώ συγγνώμη και από τους διερμηνείς, λέει η κυρία Γιάνσλοβίτσκα. Τον Μάρτιο λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, εκπώνησε ε, οδηγία για την επιβολή της οδηγίας 96-71. Μετά από 16 ε, χρόνια βεβαίως πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω η προστασία των εργαζομένων και πρέπει να έχουμε συστήματα έτσι ώστε η απόσπαση να γίνεται με τον πιο νομικό, νόμιμο συγγνώμη, τρόπο. Ε, οι εργαζόμενοι σε αυτήν την περίπτωση πολύ συχνά ε, υφίστανται περισσότερο την κρίση ε, και πολύ συχνά επίσης συμμετέχουν σε ένα είδος κοινωνικού dumping. Βεβαίως η οδηγία βασίζεται στην ε, ελεύθερη διακίνηση των αγαθών και όχι των ε, ε, ελεύθερη κυκλοφορία των ανθρώπων. Επομένως δεν καταλαβαίνουμε γιατί έπρεπε να βασιστεί στην οδηγία που αφορά τις υπηρεσίες. Ο, ο εργαζόμενος πληρώνεται στην χώρα στην οποία εργάζεται, ενώ οι εισφορές καταβάλλονται στην χώρα ε, από την οποία έχει ε, ξεκινήσει. Επομένως, δεν μπορούμε και δεν πρέπει να μιλάμε για κοινωνικό dumping ε, η απόσπαση των εργαζομένων παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο <coughs> για την ολοκλήρωση της ενιαίας ε, αγοράς ε, και βεβαίως και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, τελικά κερδίζει από την απόσπαση εργαζομένων ε, πρώτη σε αριθμό ε, από τους οποίους έρχονται οι Πολωνοί ακολουθούμενοι από τους Γάλλους και τους Γερμανούς και η ανταγωνιστικότητα ενισχύεται και το δυναμικό το οποίο μεταφέρεται είτε δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας είτε ε, ενισχύει την τοπική αγορά εργασίας. Έχουμε δει βεβαίως ότι υπάρχουν πολλές περιπτώσεις παραβίασης των ε, ε, δικαιωμάτων των εργαζομένων, όπως ας πούμε στην περίπτωση της Φλάμενβιτ οι συμβάσεις των εργαζομένων έχουν υπογραφεί για διασυνοριακή εργασία. Ε, έχουμε πάντως πολλά παραδείγματα ε, τα οποία αφορούν την παραβίαση των δικαιωμάτων εργαζομένων στα πλαίσια της απόσπασής τους. Δεν είναι πάρα πολλές ε, οι περιπτώσεις, αλλά είναι τέτοιες που μας οδηγούν σε το να υποβάλλουμε προτάσεις έτσι ώστε να αποφευχθούν τέτοιου είδους παραβιάσεις. Εγώ ασχολήθηκα κυρίως με τα θέματα τα οποία αφορούν την νομική σαφήνεια την ε, σαφήνεια ε, όσον αφορά ε, την διοικητική συνεργασία καθώς επίσης και την κινητροδότηση για τις επιχειρήσεις. συνειδητοποιήσαμε ότι τα 3, 5, 9 και 12 είναι τα άρθρα τα οποία είναι πιο προβληματικά και το κεφάλαιο 6 όσον αφορά την εφαρμογή ε, των αποφάσεων διασυνοριακά. Όσον αφορά το άρθρο 5 πρέπει να πω ότι ε, το, εδώ δεν αναφερόμαστε μονάχα στις ε, εταιρείες οι οποίες δεν ε, σέβονται τους κανόνες, αλλά υπάρχουν και αυτές οι οποίες δεν δίνουν αρκετές πληροφορίες όσον αφορά την ίδια την εργασία. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο συνήθως το ξεπερνούν όλοι πάρα πολύ εύκολα. Λέμε εμείς ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε καλύτερη πληροφόρηση, αλλά βεβαίως και όσον αφορά την ίδια την πληροφόρηση να είναι πιο αυστηροί οι κανόνες. Ε, και τελικά να αποφύγουμε τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι ε, λόγω του ότι η αγορά εργασίας δεν είναι ε, διαφανής. Προνείνω να δημιουργηθεί μία, μία και μόνη υπηρεσία πληροφόρηση σε κάθε χώρα, να υπάρχει μονάχα ένα ιστότοπος, ένα ε, ένας ιστότοπος ο οποίος αναχώρα, στον οποίο μπορεί να ανατρέξει κανείς έτσι ώστε να βρει όλες τις ε, πληροφορίες. Ε, και επίσης όλες οι αναφορές στον ιστότοπο να είναι υποχρεωτικές. Κατά την όψή μου με τον τρόπο αυτό θα υπάρξει και σαφήνεια και βεβαιότητα όσον αφορά την ε, πληροφόρηση. Γιατί μην λησμονούμε ότι κάθε χώρα έχει τις της αρχές, κάθε χώρα έχει άλλες ε, άλλου είδου ανάγκες και επομένως για τον λόγο αυτό θα πρέπει να υπάρχει μια κοινή αντιμετώπιση Εάν θέλουμε να ε, σέβονται αυτούς τους ε, κανόνες ή ε, επιχειρήσεις, θα πρέπει να διευκολύνουμε την πρόσβαση στην πληροφόρηση. Οι εργαζόμενοι, αλλά και οι χρήστες των υπηρεσιών, θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα να προστρέχουν σε με πληροφορίες τις οποίες θα βρίσκουν στα αγγλικά και στην γλώσσα της χώρας την οποία πρόκειται πρόκειται να αποσπαστούν. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία και περιέχονται στα άρθρα 3 και 9. Το άρθρο 3 προβλέπει μία σειρά στοιχείων που καθορίζουν εάν πρόκειται για πραγματική περίπτωση απόσπασης εργαζομένων. Ε, πρώτα απ' όλα θα πρέπει να αναλυθεί η δραστηριότητα της εταιρείας, της επιχείρησης και μετά η φύση του αποσπαζόμενου εργαζόμενου. Ε, όμως θεωρούμε ότι οι αναφορές εδώ δεν είναι εξαντλητικές και στις δύο, στους δύο καταλόγους ε, ανατρέχουμε γιατί δεν, έχουν σωστά, δεν έχει σωστά εφαρμοστεί ε, το δίκαιο και υπάρχουν επίσης ε, και εταιρείες οι οποίες αποκλείονται εντελώς από κάποιες αγορές και από κάποιους χώρες. Εγώ προτείνω λοιπόν να είναι ανοιχτός ο κατάλογος. Εμείς προτείνουμε μία τροποποίηση όσον αφορά ε, το 3.1α και το 3.1β, δηλαδή ε, ε, όσον αφορά τους παράγοντες των επιχειρήσεων. Εμείς θεωρούμε ότι αυτά τα στοιχεία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Επίσης να πω ότι η απόσπαση δεν είναι εθνικό φαινόμενο, είναι διασνοριακό. Γι' αυτό λοιπόν χρειαζόμαστε ένα ενιαίο νομικό πλαίσιο. Στο άρθρο 9 όμως άρθρο 9 το οποίο αφορά τους εθνικούς μηχανισμούς ε, ελέγχου. Εδώ υπάρχει ένας κατάλογος που έχει ε, εκπονήσει η Κομισιόν για τον έλεγχο των επιχειρήσεων. Ε, έχει μία σειρά εργαλείων αναφέρεται επίσης η Κομισιόν και σε μια κοινοποίηση ε, η οποία θα πρέπει να λάβει χώρα την ε, στιγμή της ε, έναρξης των εργασιών του αποσπαζόμενου εργαζόμενου. Θα πρέπει και να υπάρχει ενδεχομένω και κάποιος εκπρόσωπος των συνδικάτων εάν παραστεί ανάγκη για περαιτέρω διαπραγματεύσεις. Ε, ο κατάλογος των εργαλείων είναι κλειστών και επομένως εμείς αναφερόμαστε εδώ και σε κάποια επιπλέον στοιχεία όσον αφορά το όργανο του, του, ελέγχου. Ποιο είναι ακριβώς αυτό το όργανο του ελέγχου. Επίσης πιστεύουμε ότι θα πρέπει, μάλλον ότι είναι δυνατόν να προσθεθούν ε, κάποια κριτήρια κριτήρια επιπρόσθετα έτσι ώστε να είμαστε βέβαιοι ε, ότι δεν υπάρχει παραβίαση των δικαιωμάτων από πλευράς της επιχείρησης. Όσον αφορά τους ελέγχους, τα κράτη-μέλη τα οποία υποδέχονται ε, αποσπασμένους εργαζόμενους ε, θα πρέπει να είναι σε θέση να ελέγχει και να ε, προχωράει σε διακριβώσεις αλλά βεβαίως δεν ε, μπορεί με κανένα τρόπο να απαγορεύσει στην εταιρεία να αποσπάσει εργαζόμενους. Γι' αυτό ακριβώς εμείς λέμε ότι θα πρέπει να ε, υπάρχει το πρωτόκολλο κάθε φορά του επιθεωρητού, ο οποίος έχει κάνει την επιτόπου επιθεώρηση από την επιθεώρηση εργασίας βέβαια. Και όσον αφορά τώρα αυτούς τους ελέγχους, τις επιθεωρήσεις και τις κυρώσεις, ε, κάνουμε κάποιες ε, προτάσεις έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν ε, οι απαιτήσει των κοινωνικών εταίρων. Θέλουμε να υπάρχουν και κάποια πιστοποιητικά για τις εταιρείες οι οποίες είναι άμεμπτες και επίσης να έχουμε ένα κατάλογο των εταιριών οι οποίες δουλεύουν και σέβονται ε, όλες τις αρχές. Επίσης έχουμε το άρθρο 12, το οποίο αφορά την ευθύνη. Κοιτάξτε, εδώ γίνεται μια προσπάθεια να μην ε, ε, υπάρχει τόσο εκτενής ε, εγώ λέω ότι θα πρέπει να διαγραφεί ε, αυτό το άρθρο, διότι πιστεύω ότι οι εταιρείε οι οποίες ε, προχωράνε σε απόσπαση εργαζομένων μπορεί να δουλέψουν σε περιπτώσεις ή σε χώρες οι οποίες δεν έχουν τις ίδιες ε, υποχρεώσεις, αλλά όμως, μια και μιλάμε για διασυνοριακή ε, διαδικασία, ε, θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι είτε επιλεγεί η μεδαπός είτε αλλοδαπός συνεργάτης θα έχει ακριβώς τις ίδιες ευθύνες. Ε, και ε, επομένως για τις περιπτώσεις ε, υπεργολαδίας το να πούμε ότι θα υπάρχει από κοινού και εις η ευθύνη μπορεί να μην αναγνωρίζεται σε άλλες χώρες και θεωρούμε ότι αυτή η από κοινού και εις ευθύνη δεν βοηθάει πάντοτε τους εργαζόμενους. Εάν το άρθρο 12 θέλει πραγματικά να προστατέψει τους εργαζόμενους, στην ουσία, με το άρθρο αυτό καλύπτονται μονάχα οι αποσπασμένοι εργαζόμενοι και όχι οι ε, αυτόνομοι εργαζόμενοι, ε, δηλαδή μονάχα οι μισθωτοί αποσπασμένοι καλύπτονται. Και όχι οι ελεύθεροι επαγγελματίες ε, ή ανεξάρτητα εργαζόμενοι. Αυτό το εργαλείο της σε ολόκληρων ευθύνη θα πρέπει να αφορά και να επιβάλλεται σε όλες τις ε, εταιρείε, ε, οι οποίες θα πρέπει βεβαίως να σέβονται και την due diligence και Πρέπει μην ξεχνούμε ότι έχουν φτάσει και κάποιες υποθέσεις ε, στην, στο δικαστήριο. Εν πάση περιπτώσει, εγώ είμαι κατά της προτάσεως του άρθρου 12 έτσι όπως προτείνεται από την Κομισιόν. πρόκειται για υποχρεώσεις οι οποίες αφορούν μονάχα τις εταιρείε ε, οι οποίοι αποσπούν ε, εργαζόμενους και όχι στους άλλους, μισθωτούς τέλο πάντων. Ξέρω ότι μέσω της συζήτησης ε, θα μπορέσουμε να Ε, θα μπορέσουμε να κάνουμε και τροποποιήσεις. Ε, θα ήθελα να ασχοληθώ και με δύο άλλα σημεία. Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και εκτέλεση των αποφάσεων διασυνοριακά. Όσον αφορά τη διοικητική συνεργασία, αναφέρομαι στα άρθρα 6, 7 και 18 που αποσαφηνίζουν τους όρους της διοικητικής συνεργασίας. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπει προθεσμία 24 ώρων για τις επίγουσες περιπτώσεις και ε, προθεσμία δύο εβδομάδων για τις ε, Στάνταρτα διαδικασίες. Προτείνει επίσης να χρησιμοποιείται το σύστημα IMI για την ανταλλαγή ε, πληροφοριών μεταξύ των διαφόρων διοικητικών οργανισμών ε, των κρατών μελών. Είναι ένα εργαλείο το οποίο έχει ένα σύστημα το οποίο έχει ε, χρησιμοποιηθεί πολύ και οδηγεί σε γρήγορη ανταλλαγή ε, απόψεων. Όσον αφορά το άρθρο 18, κατά την άποψή μου, είναι πολύ γενικευτική η αναφορά στην ανταλλαγή ε, πληροφοριών όσον αφορά την απόσπαση εργαζομένων. Εγώ ε, θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχουν τρεις προθεσμίες δύο ημέρες για τις επίγουσες, δύο εβδομάδες και μήνας, ε, δύο εβδομάδες ε, για σταθερές, στάνταρ μάλλον ε, περιπτώσεις και προθεσμία ενός μήνα, σε περίπτωση κατά την οποία η πληροφόρηση απαιτεί πρώτερο έλεγχο από πλευράς των ελεγκτών. Προτείνουμε λοιπόν και την επιβολή του συστήματος, χρήσης του συστήματος IMI, οποτεδήποτε αυτό είναι δυνατόν. και να πρόκειται για σύστημα το οποίο θα πρέπει να έχει προτεραιότητα ακόμα και επί των ε, διακρατικών ε, σχέσεων. Θα ήθελα τώρα να μου πείτε, ε, αγαπητοί συνάδελφοι, ποια είναι η άποψή σας. Πώς βλέπετε το θέμα. θα ήθελα να έχουμε μια καλή συνεργασία με όλους τους συναδέλφους για να καταλάβουμε όλοι πώς λειτουργεί αυτό το σύστημα IMI. Θα έχουμε λοιπόν μια συνάντηση ε, στην οποία καλώ όλους τους ε, παρισταμένους. Θα σας καλέσω και συγκεκριμένα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Όσον αφορά τώρα την ε, εφαρμογή των αποφάσεων. Πρόκειται για ένα κεφάλαιο, είναι το κεφάλαιο 6. Το έχουμε στείλει στην Νομική Επιτροπή ε, γιατί χρειαζόμαστε γνωμοδότηση της Νομικής Επιτροπής. Φρονούμε ότι αν δεν υπάρχει ομοιογένεια ε, των ε, και των, και των αποφάσεων και των ποινών, τότε θα έχουμε πρόβλημα. Έχουμε δύο περιπτώσεις που το σύστημα δεν λειτουργεί. Ε, και ε, επομένως ε, για την ώρα δεν έχουμε ομοιομορφία αλλά χωρίς ομοιομορφία όμω δεν μπορεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο να εφαρμοστεί το σύστημα περιμένουμε όμως είμαστε σε αναμονή της απόφασης της ε, ε, Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων. 13 ε, Δεκεμβρίου προθεσμία υποβολής τροπολογιών, 23-24 Ιανουαρίου του 2013 μελέτη των τροπολογιών, μετά θα έχουμε μελέτη των συμβιβασμών στις 20 Φεβρουαρίου και τέλος ψηφοφορία την 21η Φεβρουαρίου του 2013. Και άλλη μία όμως σημαντική ημερομηνία 16 ε, Δεκεμβρίου η Έσκο θα παρουσιάσει μία έκθεση για την πρόοδο των εργασιών στο Συμβούλιο. Πρόκειται για συζήτηση προσανατολισμού, να δούμε πώς ε, προχωρούν οι συζητήσεις όσον αφορά τους αποσπασμένους εργαζόμενους. Αυτά ήθελα να σας πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Ε, και βεβαίως ε, θα πρέπει να το συζητήσουμε γιατί από ό,τι καταλαβαίνω υπάρχουν πολλές αμφισημίες ε, στην οδηγία. Εγώ προτείνω μια κανονιστική προσέγγιση στην οδηγία αυτή, συνάντηση με τους κοιόδης εισηγητές έτσι ώστε να μπορέσουμε να συζητήσουμε εντελεχέστερα την πρόταση της Κομισιόν. Αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ βεβαίω και ήδη και τους συναδέλφους που έχουν ήδη συμμετάσχει στις συζητήσει αυτές και τι συναντήσει. Ελπίζω ότι θα είναι καρποφόρο για όλους αυτή η συνεργασία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, ευχαριστώ πολύ την εισηγήτρια. Θα ήθελα απλώ να πω μερικά πράγματα για το χρονοδιάγραμμα. δεν αφορά βέβαια μόνο την έκθεση, αλλά έχει να κάνει και μια συνολική απόφαση ε, του, της Επιτροπής. Θέλω με την ησυχία μας να το συζητήσουμε αυτό το θέμα. Θα σας πω ποιος έχω συμπεριλάβει στον κατάλογο των ομιλητών για να μην υπάρχει σύγχυση. Θέλω επίσης να δώσω το λόγο και στον εισηγητή της Επιτροπής των Περιφερειών τον κύριο Χάτσινσον, ο οποίος είναι εδώ, και στον κύριο Σίλβα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Λοιπόν, σκιώδεις εισηγητές. Χιούζ, Ιρς, Σρέτερ, Χάντελ, εκ μέρους των ομάδων, Μαν, Στάινρουκ, Τούρουνεν, που είναι και η συγγήτρια για την γνωμοδότηση, συντάκτρια γνωμοδότησης για την ΙΜΚΟ, Ρέγνερ, Μπένιον και Κλωσόφσκι. Παρακαλώ, ό,τι θέλετε να πείτε να το πείτε. Μήπως ξέχασα κανέναν, θέλει κανείς άλλος να ε, πάρει το λόγο. Κύριε Όρη, κύριε Σέρκας, κύριε Μάκιντάρ. Όχι οι συντονιστές δεν θέλουν να πάρουν το λόγο μετά. Α, ναι. Ε, ξυπνήστε λοιπόν, γιατί μετά θα κλείσω τον κατάλογο των ομιλητών. Κύριε Ορή, δεν θέλετε να πάρετε το λόγο. Ε, εντάξει, αφού δεν θέλετε. Μάκινταρ και Σέρκας λοιπόν προσθέτω στον κατάλογο των ομιλητών και κλείνω τον κατάλογο των ομιλητών. Στίβεν Χιούς πρώτος. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ την εισηγήτρια. Είχαμε συναντηθεί, ξέρει ότι σε μερικά σημεία διαφωνούμε. Ε, μάλιστα συμφωνούμε σημαντικά σε μερικές σημαντικές πτυχές της οδηγίας αλλά τέλος πάντων υπάρχει ένα πράγμα επί το οποίο συμφωνούμε μέγιστη νομική σαφήνεια στο κείμενο που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν δίνει την ε, απαραίτητη νομική σαφήνεια, οπότε πρέπει να περάσουμε στη διαδικασία των τροπολογιών και στη συζήτηση βέβαια για να βελτιώσουμε το κείμενο της Επιτροπής. Υπάρχουν ε, ιδιαίτερε ευαισθησίε γύρω από αυτό το θέμα, το γνωρίζετε. Η εισηγήτρια μάλιστα αναφέρθηκε στην πρώτη τη τροπολογία όταν άρχισε την παρέμβασή τη και νομίζω ότι ευθύ εξ αρχή πρέπει να πούμε ότι αυτέ οι ευαισθησίε ε, κάπω επειδή έχουμε αυτές τις συζητήσεις, ε, ε, έχουμε αυτές τις συζητήσεις επειδή υπήρξαν ε, κάποιες αποφάσεις του δικαστηρίου πριν από μερικά χρόνια. Θα θυμάστε τι σημαίνει αυτό, τι σημαίνει αυτό περί τίνος το τέλος πάντων αφορούσε από τη μία το δικαστήριο έπρεπε να ασχοληθεί με την ελευθερία των εργαζομένων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την άλλη ελευθερία παροχής διασυνοριακών υπηρεσιών που είχαν το πάνω χέρι. Και το γεγονός ότι επιλήφθηκε το δικαστήριο δημιούργησε κάποια ε, φιλονικία. Στη δεύτερη αιτιολογική σκέψη λοιπόν η εισηγήτρια θεωρεί ότι η ελευθερία παροχής υπηρεσιών είναι βασική προτεραιότητα ενώ το κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θεωρεί πρωταρχική προτεραιότητα τη μετακίνηση των εργαζομένων. Έχουμε μακρύ κατάλογο μιλητών, οπότε θα προσπαθήσω να βασιστώ στι κύριε πτυχέ διαφωνία, αλλά ούτω ή άλλω θα χρειαστεί να γεφυρώσουμε τι διαφορέ μα εδώ στην Επιτροπή. Άρθρο 2 για του ορισμού. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό στην παράγραφο D του 2 όταν ορίζουμε την διακρατική παροχή υπηρεσιών πρέπει να το ορίσουμε σαφώς ε, βάσει των άρθρων 15 και 49 των συνθήκων. Αυτό είναι κάτι ε, επί του οποίου θα τροπολογήσω. Δεύτερον, ε, μία νέα παράγραφο ΣΕΦ στο άρθρο 2 θα μπορούσε να, αφορά, να χρησιμοποιεί τη διατύπωση από την αρχική οδηγία 96 για τον ορισμό τι είναι το κράτος υποδοχής θα ήθελα και πάλι να υπάρχει, μια, να υπάρχει επαρκή σαφήνεια για το θέμα αυτό. Χρειαζόμαστε επίσης και ένα νέο άρθρο 3 για το πεδίο εφαρμογή της οδηγίας. Ε, θέλουμε νομίζω να ε, δούμε τι σχέση υπάρχει μεταξύ της οδηγίας των αποσπασμένων αλλά και των εποχιακά εργαζόμενων ε, βάσει της οδηγίας ε, της αρχικής του 96 υπό το φως των απαιτήσεων των προσωρινών για σαφείς διατάξεις ισότητας. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό ε, πρέπει να το συμπεριλάβουμε. Επίσης πρέπει να αναφέρουμε σαφώς ε, αυτή η οδηγία επιβολής κατά πόσο θα ισχύει για υπηκόους τρίτων χωρών. Για το άρθρο 3 τώρα, για τα στοιχεία εφαρμογής και παρακολούθησης, εμείς θα θέλαμε να υπάρχουν κάποια κριτήρια που δεν θα είναι διεξοδικά που είναι κάτι το αντίθετο βέβαια από την άποψη της εισηγήτριας. Θα θέλαμε να συμπεριλάβουμε σημεία στον κατάλογο. Η εισηγήτρια είπε ότι συμφωνεί να συμπεριληφθούν νέα σημεία. Κάτι το οποίο θα ήθελα να προτείνω εγώ είναι η αναφορά στο, στο ποσοστό ε, συμμετοχής ε, ε, της ε, χώρας προέλευσης Νομίζω ότι τα περαιτέρω μπορούμε να τα δούμε αργότερα. Στο άρθρο 3, παράγραφος 2, εκεί που λέει κατά πόσο ένας προσωρινά εργαζόμενος έχει ε, καθήκοντα και σε κάποια άλλη χώρα, ε, νομίζω ότι δεν πρέπει να είναι διεξοδικός ο κατάλογος αυτός. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Επίσης, θα θέλαμε να προσθέσουμε θα πρέπει να προσθέσουμε και κάτι άλλο σε αυτό το τμήμα του κειμένου λέει ότι εάν ο εργαζόμενος ε, δεν, εάν ο εργαζόμενος δεν μπορεί να πει ότι εργάζεται σε μια άλλη χώρα από αυτήν που ισχυρίζεται ότι εργάζεται, τότε θα θεωρηθεί ότι η σχέση εργασίας θα διέπεται από το κράτος εργασίας ε, στο οποίο ε, ε, γίνεται η εργασία. Προσπαθώ να τα πω αργά, λέει ο κύριος Χιούς πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, γιατί αν δεν είμαστε προσεκτικοί μπορεί να ε, μην συνάδουμε με τη Ρώμη 1 στη συγκεκριμένη διατύπωση. Γιατί αν δεν το κάνουμε αυτό θα διέπεται από τη Ρώμη 1, οπότε μπορεί η χώρα προέλευσης να είναι ε, η χώρα της, ε, της οποίας το, το δίκαιο θα υπερέχει. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί ως προς αυτό. Χρειαζόμαστε και ένα νέο άρθρο 3, παράγραφος 3, ένα νέο κατάλογο κριτηρίων ε, για τον ορισμό του κατά πόσο ένα άνθρωπο είναι αυτοαπασχολούμενο ή όχι στη χώρα υποδοχή. Η συγκήτρια αναφέρθηκε στο γεγονό ότι ένα από του τομεί όπου ε, γίνονται καταχρήσει και νομίζω ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να το τονίσουμε αυτό και να το ε, να το διευκρινίσουμε στο κείμενο. Ένα άρθρο 4 θα αναφέρει τον κατάλογο των δικαιωμάτων των ε, εργαζομένων, ε, δηλαδή στέγαση, να εξασφαλίζεται δηλαδή ότι υπάρχουν, ε, ότι εξασφαλίζονται τα δικαιώματα των αποσπασμένων. Για το άρθρο 7 έχουμε ίσονο σημασία τροπολογίε. δεν έχω τίποτε το ιδιαίτερο να πω από πλευρά σοσιαλδημοκρατών. Το άρθρο 9 όμω για τα εθνικά μέτρα ελέγχου, νομίζω ότι πρέπει να είναι σαφές ε, ότι ο κατάλογος των διοικητικών απαιτήσεων και ελεγκτικών μέτρων δεν θα είναι προαιρετικός. Πρέπει να το διευκρινίσουμε αυτό, ότι αυτά, αυτοί οι διοικητικές απαιτήσει και τα μέτρα ελέγχου θα επιβάλλονται, σαλ δηλαδή πρέπει να γράψουμε, και τελευταίο θα ήθελα να αναφέρω το άρθρο 12 για την κοινή ευθύνη. Σε κάποιο βαθμό έχει άμεση σχέση και με τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών ε, για την ε, εφαρμογή της ε, οδηγίας του 96. Έδωσα στην εισηγήτρια ένα αντίγραφο της ανταλλαγής αλληλογραφίας που είχα με το GNB, το δικό μου το συνδικάτο, και αφορά την υπεργολαβία για ε, ένα έργο στην βορειοδυτική Αγγλία, τη Siemens, όπου 14 Πολωνοί εργαζόμενοι ε, έχουν προσληφθεί και δεν έλαβαν την αποζημίωση ε, την οποία έπρεπε να λάβουν. Το συνδικάτο έλαβε, ανέλαβε δράση και πήραν μια αποζημίωση 270.000 λιρών. Ε, όμως ε, η συγκεκριμένο υπεργολάβος γύρισε πίσω στη χώρα του και υπήρχε πολύ μεγάλο πρόβλημα με το να τους βρούμε. Ρωτήσαμε τη Siemens, η Siemens μας είπε δεν μπορεί να βοηθήσει, δεν ξέρει τι έγινε αυτός ο υπεργολάβος που χάθηκε, παρά το γεγονός ότι κανονικά θα πρέπει να έχουν κάποιο γραπτό αρχείο από πού ήρθε αυτός ο υπεργολάβος στο Αμβούργο έγραψε ε, ο υπεργολάβος, γράψαμε σε έναν υπεργολάβο που θεωρούσαμε ότι είναι στο Αμβούργο, αλλά τελικά εκείνοι μας απάντησαν, απάντησαν ότι όχι, δεν έγινε κάτι τέτοιο, δεν είμαστε εμείς ο υπεργολάβος. Τέλο πάντων, υπήρχε μια τεράστια σύγχυση. Τέτοιου είδου προβλήματα πρέπει να τα αποφύγουμε ή τέλο πάντων να προσπαθήσουμε. Ένα συνάδελφο αναφέρθηκε στο Φλάμονβιλ, ένα παράδειγμα ακραίο του πόσο μπορούν να πάνε στραβά τα πράγματα, συνεργασία, υπεργολαβίε ε, κλπ. Έχουμε τέτοιου είδους παραδείγματα ενός υπεργολάβου ο οποίος εξαφανίζεται και δεν σέβεται τις υποχρεώσεις του. Ε, μερικές φορές μάλιστα υποχρεώσεις ε, οι οποίες ε, έχουν επιβληθεί από τα δικαστήρια. Εμείς πιστεύουμε λοιπόν ότι χρειάζεται ένα άρθρο 12 για την κοινή ευθύνη παρόλο που η συγχύτρια λέει ότι δεν θα έπρεπε να είναι εκεί αυτό το άρθρο. Διαφωνούμε λοιπόν με πολλούς τομεί. Ε, μπορούμε να γεφυρώσουμε κάποιες από τι διαφορές μας και να συνεργαστούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Η συγχύτρια είπε ότι θα το κάνει αυτό, θα κάνουμε κι εμεί ό,τι μπορούμε για να ε, την συναντήσουμε κι εμεί κάπου στη μέση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νάντια Ήρς και μετά Σρέτερ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω καταρχάς την εισηγήτρια για την εξαιρετική και πολυκοπιαστική δουλειά που έκανα μαζί και με τους σκιώδεις εισηγητές. Το σχέδιο που έχουμε εδώ έχει ορισμένες ε, καλές αφετηρίες, όμως για μας ορισμένα σημεία φτάνουν πολύ ε, πέραν των αρμοδιοντήτων τους και άλλα όχι αρκετά όσο θα τα θέλαμε. Καταρχάς άρθρο 5. Εδώ πιστεύω σίγουρα πώς θα μπορούσαμε να σκεφτούμε να υπάρξει και μια ιστοσελίδα για τα κράτη-μέλη που μπορούν να βρουν πληροφορίες. Θα ήταν μια καλή ε, έτσι, προσέγγιση όπου οι πληροφορίες θα μπορούσαν να είναι στα αγγλικά. Όμως εδώ βρίσκουμε μια δυναμία στη διατύπωση προς το παρόν ε, αναφέρεται στις σημαντικότερες άλλες γλώσσες. Και μπορεί να ρωτήσει κανείς και καλά θα κάνει ποιες είναι οι άλλες σημαντικές γλώσσες. Είναι πολύ σημαντικό για μας από τη μία η χώρα υποδοχής να, έχει, να χρησιμοποιεί και την γλώσσα, αλλά να χρησιμοποιείται επίσης και η γλώσσα της χώρας προέλευσης του εργαζομένου. Δηλαδή, όταν ένας ε, Ούγγρο ε, εργαζόμενο, δουλεύει για μια πολωνική εταιρεία και πηγαίνει στο Ηνωμένο Βασίλειο, πρέπει οι πληροφορίε να υπάρχουν και στα ουγγρικά. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό οι πληροφορίε να βρίσκονται στη διάθεσή του στην γλώσσα του, στην γλώσσα τη χώρα προέλευση. Τώρα, άρθρο 3.9 για τις δυνατότητες ελέγχου και την συζήτηση για την ε, κλειστή ή ανοιχτή λίστα. Ε, λοιπόν, πιστεύω ότι από τη μία μπορούμε να κατανοήσουμε ότι η κλειστή λίστα είναι συνετή για λόγους ε, ασφαλείας. Ωστόσο, εδώ υπάρχουν ένα, κάποια σημεία τα οποία χρειάζονται προσθήκες, διότι για εμάς ε, μία λίστα που θα μας δίνει δυνατότητες ελέγχου χρειάζεται. Η άλλη επιλογή θα ήταν μια ανοιχτή λίστα, όμως εκεί το πρόβλημα που υπάρχει είναι το τι θα περιέχει αυτή η λίστα και είμαι σίγουρη όμως ότι θα καταλήξουμε σε μια συμβιβαστική λύση. Μετά ή τώρα, γενικά, σε γενικές γραμμές, για το άρθρο 12, πιστεύω ότι η διαγραφή ίσως είναι υπερβολική. Ίσως εμείς θα έπρεπε να αναλογιστούμε για το ποιος είναι ο στόχος μας. Και ποιος είναι ο στόχος μας. Ο στόχος μας είναι οι εργαζόμενοι να πάρουν την αμοιβή τους, αλλά και τις ε, εισφορές τους για την κοινωνική ασφάλιση και να, και εκπληρώσουν τις ε, δικές τους υποχρεώσεις για τη φορολογία, για παράδειγμα. Έχουμε πολλά διαφορετικά τέτοια συστήματα στα κράτη-μέλη, ορισμένα δεν έχουν κανένα, ορισμένα έχουν παραβι... σε ορισμένα παραβιούνται παραβιάσεις. Στη Γερμανία υπάρχει η ευθύνη για το χρέο, αλλά πιστεύω ότι σε γενικέ γραμμέ δεν πρέπει να χάσουμε από τα μάτια μας το στόχο. Δηλαδή, να ανοίξουμε το δρόμο για τα κράτη-μέλη και να τους δώσουμε μια ξεκάθαρη διατύπωση εδώ για το άρθρο 12, όπου να αναφέρεται ρητά η περιγραφή του μισθού, των απολαβών, των κοινων... της κοινωνικής ασφάλισης, της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Ίσως εδώ θα μπορούσαμε να ε, παραπέμψουμε σε μια άλλη οδηγία στην Οδηγία 2009 κάθετος 52 που αναφέρεται στην, ε, μαύρη, στην παράνομη εργασία και εδώ αναφέρονται και οι μετανάστες. Και θα μπορούσαμε να κοιτάξουμε αυτήν την οδηγία για να δούμε πώς θα πετύχουμε το στόχο μας, πώς δηλαδή οι εργαζόμενοι θα πάρουν τις απολαυές τους και τα υπόλοιπα ε, που δικαιούνται. Ίσως δηλαδή εδώ να μπορούσαμε να βρούμε ένα συμβιβασμό για την μέθοδο που θα ακολουθήσουμε για να φτάσουμε στο στόχο μας. Πιστεύω πως ε, γενικά το θέμα είναι πάρα πολύ δύσκολο και μεγάλο, το ξέρετε όλοι, αλλά έχουμε μια δυνατότητα εδώ να βρούμε μια καλή λύση. Ευχαριστώ. Elizabeth puis Thomas. Ε, Elizabeth και μετά Thomas Handel. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχά να ευχαριστήσω και εγώ την εισηγήτρια για την παρουσίαση. Ήταν μακροσκελέστατη παρουσίαση, περάσαμε πάρα πολύ καιρό συζητώντα το θέμα και, το πιστεύω, και πιστεύω πως αυτό ήταν καλό, διότι έτσι μπορούσαμε να εμβαθύνουμε. Για μένα, που ασχολήθηκα πάρα πολύ με αυτό το φάκελο, μία από τις, ε, μία, ένα από τα κεντρικότερα ερωτήματα είναι η σχέση με την παλαιότερη οδηγία, με την ισχύουσα οδηγία και εδώ ίσως πιστεύω πως είναι σημαντικό να δούμε εάν θα πρέπει να αλλάξει αυτή η οδηγία, διότι τι θα κάνουμε, είναι καλύτερο να αλλάξουμε την ισχύουσα οδηγία ή να εφαρμόσουμε αυτά που μας προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με έμεσο τρόπο και εμείς είμαστε, έχουμε ξεκαθαρίσει θέση. Πιστεύουμε ότι όλα τα πράγματα που είναι σημαντικά και περιέχονται σε αυτή την οδηγία πρέπει να είναι και η βάση μας, η βάση την οποία θα ακολουθήσουμε. Δηλαδή η τωρινή ισχύουσα οδηγία, η οδηγία εφαρμογής πρέπει να έχει ως στόχο να βελτιώσει τις πρακτικές, να βελτιώσει αυτό που γίνεται τώρα και όχι να δημιουργήσει καινούρια νομική βάση. Κάτι άλλο που θα το ξέρει και όποιος ασχολείται με το θέμα. Ο Στίβεν Χιούς ίσως το ανέφερε. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά το ρόλο των κρατών μελών στα οποία λαμβάνει η χώρα η εργασία έχει καθοριστεί εκ νέου. Και κάποια άλλα κράτη-μέλη στα οποία αποσπώνται οι εργαζόμενοι <clears throat> αναφέρονται Εκ ναι, Όμως με αυτό το θέμα ασχολείται η Οδηγία για την παροχή υπηρεσιών και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να προσπαθήσουμε όχι να βελτιώσουμε το πώς γίνεται αλλά να το επαναλάβουμε. Αλλά δεν θέλουμε να επαναλάβουμε αυτά που έχουν ήδη υποθεί. Σίγουρα αυτό δεν χρειάζεται να το εξηγήσω σε όσους ξέρουν την ιστορία λίγο καλύτερα. Αλλά να πω ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, διότι ο στόχος μας είναι ο ρόλος των κρατών μελών στα οποία λαμβάνει η χώρα εργασία να ενισχυθεί και να βελτιωθούν οι πρακτικές. Αυτός είναι ο στόχος μας διότι έτσι θα είμαστε και συνεκτικοί ως κοινοβούλιο. Τώρα, όσον αφορά τα, τις μεθόδους ελέγχου από ε, τα κρατη συνάδελφοι που ασχολούνται χρόνια με αυτό το θέμα και έχουν μεγάλη εμπειρία μας λένε ότι το α και το ω είναι τα μέτρα ελέγχου και πολύ σημαντικό είναι να κλείσουν τα παραθυράκια που υπάρχουν ανοιχτά. Ο στόχος μας λοιπόν είναι να κλείσουν τα παραθυράκια. Και πώς θα το κάνουμε αυτό με κλειστές λίστες. Δεν γίνεται. Είναι τελείως απομακρυσμένο από οποιαδήποτε πραγματικότητα. Η δυνατότητα που θα έχουν τα κράτη-μέλη για αριθμιστικά και ελεκτικά μέτρα διατυπώνεται σαφέστατα στην οδηγία. Πρέπει να είναι δηλαδή ευέλικτα. Είναι η μοναδική δυνατότητα που έχουν. Διαφορετικά, δεν θα μπορέσουμε να πετύχουμε το στόχο μας, να βελτιώσουμε την πρακτική. Στο άρθρο 3 της αρχικής οδηγίας που αναφέρεται στο δίκαιο, στις δίκαιες απολαύες, στο δίκαιο μισθό. Και εδώ διαφαίνεται και το πρόβλημα που υπάρχει στο εργατικό δίκαιο. Και γι' αυτό θεωρώ πως είναι ενδιαφέρον, ε, για παράδειγμα στον κατασκευαστικό τομέα, και οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι να καταλήξουν σε μια κοινή θέση για αυτή την οδηγία, η οποία θα είναι ένας δίκαιος ανταγωνισμός και δίκαιες απολαμβές. Και τώρα θα περάσω σε κάποια άλλα σημεία, τα οποία για μένα είναι καλές πρακτικές δεν πρέπει να αμφισβητηθούν σε καμία περίπτωση από αυτή την οδηγία, διότι οι εμπειρίες που έχουμε από τα κράτη-μέλη είναι καλές. Καταρχάς, <clears throat> να πω επίσης ότι είναι παράδειγμα προς μίμηση καλών πρακτικών. Εδώ και, πο και εδώ και πολλά χρόνια καλούμε τα κράτη-μέλη να υπογράψουν αυτές τις συμβάσεις εργασίας. Και πιστεύω πως θα ήταν και λογικό να το ενσωματώσουμε αυτό στην οδηγία. Το ερώτημα είναι πώς θα το κάνουμε αυτό, αλλά τουλάχιστον πρέπει να φροντίσουμε αυτές οι καλές πρακτικές να μπορούν να εφαρμόζονται και να μπορούν και τα άλλα κράτη-μέλη να δίνουν διδάγματα από αυτό. Έπειτα, η πληροφόρηση των εργαζομένων και η συμβουλευτική. Αυτό εμείς το υποστηρίζουμε. Στην έκθεσή μου Είχα ήδη αναφερθεί σε αυτό, σε άλλο πλαίσιο βέβαια, σε άλλη συζήτηση, αλλά το Κοινοβούλιο ήδη έχει είχε αποφασίσει ότι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό συστατικό στοιχείο, διότι έτσι με λίγο, με λίγο κόστος μπορούμε να καταφέρουμε πάρα πολλά πράγματα. Και αυτός ο τομέας για μένα είναι κέριος έτσι ώστε να κλείσουμε αυτά τα παραθυράκια που υπάρχουν. Το τρίτο θέμα είναι το άρθρο 12. Και είναι πολύ ενδιαφέρον ε, το γεγονός ότι στα κράτη-μέλη στα οποία υπάρχει αυτή η ευθύνη δεν υπάρχει ένα αντίστοιχο άρθρο 12, διότι αυτό αναφέρεται και καλύπτεται από τις καλές πρακτικές και είναι εξαίσιο αυτό. Και έτσι πρέπει να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας, να πούμε ότι, ε, ότι θα πρέπει να εδρεωθούν οι καλές πρακτικές και να διευρυθούν και να επεκταθούν και στα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Δεν λέω ότι θα είναι εύκολο, σε καμία περίπτωση. Όμως, είναι δίκαιο, είναι ευρωπαϊκό δίκαιο και πρέπει να εφαρμοστεί. Και τώρα ολοκληρώνω για τις προθεσμίες τις οποίες μας ε, είπε η συγγήτρια. Από την εμπειρία μου και το τελευταίο πράγμα που θα πω αυτό είναι ότι οι προθεσμίε δεν είναι ρεαλιστικέ. Θέλουμε τελείω διαφορετικέ ε, προθεσμίε. Εάν πραγματικά αυτέ είναι οι προθεσμίε που προτείνετε και θέλετε να συνεργαστούμε καλά και να γίνει καλή δουλειά και, ε, στα κράτη, και ανάμεσα στα κράτη-μέλη, τότε πρέπει να αλλάξουν πολλά πράγματα. Χρειαζόμαστε πολύ μικρότερες προθεσμίες Αυτά προς το παρόν. Πιστεύω πως είμαστε ακόμα στην αρχή της συζήτησης και πραγματικά έχω μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσω τη συνέχεια. Ευχαριστώ. Ε, Δυστυχώ, ο Τόμα Χάντελ αναγκάστηκε να αποχωρήσει. Οπότε δίνω το λόγο στον Τόμας Μαν και μετά στη Γιούτα Στάιν. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και τους συναδέλφους και την εισηγήτρια. Πιστεύω πως έχετε αναφέρει πάρα πολλά σημαντικά πράγματα, μπορούμε να τα στηρίξουμε. Περισσότερη πληροφόρηση, διαφάνεια, καθα... Ε, διαφάνεια στην ανταγωνιστικότητα. Το προσυπογράφω και εγώ όλα αυτά που λέτε και περισσότερη νομική ασφάλεια. Πιστεύω βέβαια και το έγραψα και ήδη στα αγγλικά ότι για να μπορέσουμε να έχουμε μια καλή συζήτηση πρέπει να υπάρχει μια έκθεση ισορροπημένη και όχι να λέμε ότι οι επιχειρήσεις έχουν ένα πλεονέκτημα στις ε, χώρες τις οποίες προσφέρουν θέσεις εργασίας. Πρέπει να υπάρξει αυτή η καλή ε, ισορροπία και δεν πρέπει να σκεφτόμαστε με νέα κρατημέλη, παλιά κρατημέλη. Όχι. Θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό, σημαντική την προστασία των εργαζομένων. Ανεξάρτητα από το ποια ε, χώρα βρίσκονται, αν έχουν αποσπαστεί ή όχι. Πρέπει οι κανόνες να είναι σεβαστοί, όπου και αν είναι αυτό. Και ο Steve Hughes μας ανέφερε κάτι πάρα, ε, κάτι πάρα πολύ σωστό όταν ε, μίλησε και θεωρώ πως η προστασία των εργαζομένων μπορεί να είναι αποτελεσματική μόνο εάν έχουμε μια ξεκάθαρη οδηγία. Εάν ξέρουμε τι κάνουμε για να καταφέρουμε μια δίκαιη εργασία, δίκαιες συνθήκες εργασίας να αποφύγουμε επισφαλείς ε, συνθήκες ε, ε, εργασίας, επισφαλείς, συμβάσεις, προστασία, περίθαλψη. Πρέπει να διασφαλίσουμε, να ξεκαθαρίσουμε ότι οι εργοδότες θα υπόκεινται σε έλεγχο. Και εμεί έχουμε εμπειρία ε, σε, αυτό το θέμα εδώ στην Επιτροπή. Έχουμε διεξάγει θεσπέσει συζητήσει στην, ε, Επι, στην ε, Επιτροπή και με τον αρμόδιο επίτροπο. Ποιος, πρέπει να δούμε ποιος έχει δικαίωμα στα προνόμια και στις απολαβές και ποιος όχι. Δηλαδή ποιος δουλεύει νόμιμα ή όχι. Και αυτό έχει άμεση σχέση και με την κινητικότητα των εργαζομένων υπήρξαν ορισμένοι που είπαν ότι ο Επίτροπο είχε δίκιο από τα νέα κράτη-μέλη. Έχω μιλήσει με τρει συναδέλφου που βρίσκονται ακόμα εδώ στο Κοινοβούλιο, όχι σε αυτή την Επιτροπή τώρα, οι οποίοι μου είπαν ότι τώρα έχουν αλλάξει τα πάντα. Και ότι πλέον οι, εργα... οι εργαζόμενοι σε κατασκευαστικά έργα δεν είναι από τα κράτη-μέλη, αλλά είναι από τρίτες χώρε, από το Βιετνάμ, την Καμπότζη, αλλού. Και Άλλο, επίσης, είπατε ότι δεν θέλουμε εταιρείε που υπάρχουν μόνο κατ' όνομα και έχουν μια ταχυδρομική θηρίδα. Φυσικά και όχι, αλλά πώ θα το κάνουμε αυτό. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε την διατύπωση και να θεσπίσουμε ξεκάθαρα μέτρα ελέγχου. Δεν μπορώ να το τονίσω αρκετά. Μετά. Μα είπατε για τα μέτρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εδώ πιστεύω πως είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο, ένα πολύ δύσκολο τομέα. Η πραγματικότητα είναι αυτό που πρέπει να μας απασχολήσει. Υπάρχουν εθνικά μέτρα ελέγχου, πρέπει να τα, να τα χρησιμοποιήσουμε και να τα τροποποιήσουμε. Υπάρχουν ανάγκες οι οποίες μεταβάλλονται και πρέπει να προσαρμοζόμαστε σε αυτές. Τώρα, όσον αφορά και το άρθρο 12 και την ευχήνη των εργοδοτών, πιστεύω ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό για μένα δεν πρέπει να διαγραφεί, πρέπει να παραμείνει. Χρειαζόμαστε αυτούς τους προστατευτικούς μηχανισμούς σε κάθε περίπτωση. Και τέλος, θεωρώ σημαντικό και πάντα θα θεωρώ σημαντικό, διότι εμείς εδώ κάνουμε πολιτική στην Ευρώπη, ότι πρέπει η θέση των κοινωνικών εταίρων να είναι ισχυρότερη. Και εδώ έχουμε μια κοινή θέση, αλλά οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι από την εμπειρία μου πρέπει να καταλήξουν σε μια κοινή θέση. Τέλος θα ήθελα να πω ότι ελπίζω σε μια ισορροπημένη έκθεση, αλλά σας παρακαλώ μην ξεχνάτε ποτέ ότι το, οι αναγκαίες αλλαγές πρέπει να προσαρμόζονται στις αλλαγές της πραγματικότητας και να προσαρμόζονται στις θέσεις εργασίας. πρέπει να δούμε τι μπορούμε να αλλάξουμε, πότε μπορούμε να το αλλάξουμε και πώς. Αυτά από μένα. Αναμένω με αγωνία τις επόμενες συζητήσεις. Alors, euh, Steinruck, puis... Euh, Steinruck και μετά Emily Turunen. Μάλιστα. Ο στόχος μας, ο απότερος στόχος είναι η κινητικότητα και πώς αυτή θα είναι δίκαιοι. Έχουν μιλήσει πάρα πολλοί Γερμανοί ευρωβουλευτέ και αυτό πιστεύω ότι δείχνει πόσο σημαντικό είναι για εμά στη Γερμανία να υπάρχει κινητικότητα χωρίς σύνορα στην Ευρώπη και αυτό είναι σημαντικό. Σημαντικό και αναγκαίο για όλες τις χώρες και τις χώρε προέλευση και τις χώρες υποδοχής. Η Ελίζα Πεθυσχόντα το είπε ήδη. Έχουμε μια οδηγία, μια ισχυούσα οδηγία όπου παρατηρούμε ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα που χρήζουν βελτίωσης, μεγίστης βελτίωσης. Και εγώ χαίρομαι για τις συζητήσεις, αλλά να πω ότι έχετε την δυνατότητα να ασχοληθείτε με τα προβλήματα, με τα υπαρκτά προβλήματα των εργαζομένων. Εντάξει και οι εργοδότες είναι σημαντικοί, όμως οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι στο προσκήνιο. Για μένα, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η έκθεσή σας μας δίνει την δυνατότητα να ασχοληθούμε με αυτή την παραβίαση των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Το θέμα με τις εταιρείε που υπάρχουν μόνο σαν ταχυδρομική θηρίδα και με τους ελεύθερους εισαγωγικά επαγγελματίες είναι πάρα πολύ σημαντικό και πραγματικά πρέπει να το καταπολεμήσουμε. Μπορώ να σας αναφέρω παραδείγματα, 50 παραδείγματα ε, των εργασιακών δικαιωμάτων με τέτοιον τρόπο στην Ευρώπη. Είμαι κατά των, της κλειστής λίστας που αναφέρεται στο άρθρο 3 ή πρέπει να τεθούν περισσότερα κριτήρια διότι διαφορετικά μας λείπουν μας λείπει αναφορά στις συνέπειε. Τι θα γίνει δηλαδή εάν εφαρμοστούν ή όχι αυτά τα κριτήρια. Μετά αναφέρατε την πληροφορία. Είναι απίστευτα σημαντικό οι εργαζόμενοι να μπορούν να πληροφορούνται στην μητρική τους γλώσσα. Ξέρω πολλούς ανθρώπους, άριστα καταρτισμένους, οι οποίοι έχουν αυτό το πρόβλημα. Και επίσης να αναλογιστούμε σε ποιους απευθυνόμαστε και πώς θα δώσουμε τις πληροφορίες. Το ίντερνετ είναι, μια, είναι ένα πάρα πολύ καλό εργαλείο, γιατί αυτό θα μπορούσε να είναι άμεσα προσβάσιμο από οπουδήποτε και αν βρίσκεται ε, κανείς. Μετά, η ευθύνη, και αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Και πάλι έχω να σας δώσω τόσα παραδείγματα στην Ευρώπη, όχι μόνο στον κατασκευαστικό τομέα, αλλά και αλλού, όπου παρατηρούνται τεράστια προβλήματα με την εταιρική ευθύνη και αυτό που μας περιγράφει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πολύ πιο αδύναμο από αυτό που επιθυμούμε εμείς ή από αυτό που για παράδειγμα ισχύει στην Γερμανία. Χρειαζόμαστε ξεκάθαρους ορισμούς στην έκθεση με, που να αναφέρονται σε ελάχιστα, ελάχιστα στοιχεία, να τεθούν εθνικές πρακτικές για να μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Και όσον αφορά το άρθρο 9 και τα δικαιώματα ελέγχου και με τους ε, καταλόγους ανοιχτούς ή κλειστούς πρέπει τα κράτη-μέλη να έχουν τη δυνατότητα να αποφασίσουν μόνα τους για περαιτέρω ε, ελέγχους εάν θέλουν. Και τέλος να ρωτήσω την εισηγήτρια η κατάσταση τώρα στα κράτη-μέλη όπου υπάρχει ανεπαρκής έλεγχος για την, στην απόσπαση εργαζομένων. Εσείς τι προτίθεστε να κάνετε γι' αυτό. Το 2011 στη Γερμανία τα εισοδήματα από τη μαύρη εργασία ανέρχονταν στα 660 εκατομμύρια ευρώ. Γι' αυτό καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι να ελαχιστοποιήσουμε την μαύρη εργασία και επίσης να καταπολεμήσουμε την εκμετάλλευση των εργαζομένων. Διότι εάν το κάνουμε αυτό, τότε θα δημιουργήσουμε ένα καλό πρότυπο, ένα καλό επιχειρηματικό μοντέλο. Αν το αφήσουμε έτσι όμως, τότε θα συμβεί το ακριβώ αντίθετο. Ευχαριστώ. Um, Η κυρία Τούρουνεν, εγώ είμαι η συγγήτρια της γνωμοδότησης της ΙΜΚΟ, την οποία θα υποβάλουμε, την επεξεργαζόμαστε αυτή τη στιγμή στην ΙΜΚΟ. Είχαμε την πρώτη μας ε, συζήτηση για τις τροπολογίες σήμερα. Έχει γίνει λοιπόν η έκθεσή μου, υπάρχουν ήδη τροπολογίες και θα προσπαθήσω λίγο να σας πω ορισμένε ε, πτυχές από την πλευρά της Επιτροπής ΙΜΚΟ. Νομίζω ότι για όλους μας ο στόχος θα έπρεπε να είναι ε, ένα ισότιμο πεδίο και την ισότιμη προστασία των εργαζομένων, να, υπερβα, να υπερβούμε λιγάκι τα στενά εθνικά συμφέροντα. <laughs> Αφήστε το, το, το Συμβούλιο να το κάνει αυτό. Εμείς είμαστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι μακροπρόθεσμα θα έχουμε ένα ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού και ίση προστασία για τους εργαζομένους από όπου και αν προέρχονται. Αυτό είναι το ε, αυτή είναι η ανησυχία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ε, τώρα αν θέλουμε να έχουμε ένα χαμηλού κόστους, χαμηλής αποζημίωσης, ε, εργατικό δυναμικό με κακή προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων, νομίζω ότι δεν θα ευνοήσει κανέναν, ούτε την κοινωνία, ούτε την οικονομία και... Ε, θα έπρεπε να πάμε πίσω στην έκθεση Μόντι 2. Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα ε, και πρέπει να ασχοληθούμε με αυτά τα προβλήματα, να τα επιλύσουμε και να εξασφαλίσουμε ότι το ευρωπαϊκό ε, όραμα θα έχει την υποστήριξη και των εργαζομένων στο μέλλον. Και εμεί στο Ιστινίμκο τα άρθρα 3, 6, 9 και 12 θεωρήσαμε ότι είναι τα ε, πιο δύσκολα για το άρθρο 3. την πρόληψη των καταχρήσεων θα μπορούσαμε να, έχουμε έναν κατάλογο, ο οποίος όμως δεν θα είναι διεξοδικός. Για την άρθρο 6 έχουμε μια πολύ πραγματιστική προσέγγιση, ρεαλιστική σε σχέση με τις προθεσμίες. Θεωρούμε ότι είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα προς τα εμπρός και λέμε τα κράτη-μέλη που δεν συνεργάζονται να τα αναφέρουμε. Να τα αναφέρουμε, να τα δείχνουμε με το δάχτυλο. Για το 9 φαίνεται ότι μάλλον υπάρχει πλειοψηφία, αλλά είμαι μάλλον επιφυλακτική στο να το πω με βεβαιότητα, για μία ανοιχτή λίστα. Πρέπει να το συζητήσουμε περαιτέρω, όμω δεν έγινε ακόμα συνάντηση των σκιωδών εισηγητών και δεν μπορώ να το πω με βεβαιότητα. Είναι όμω ε, χρήσιμο να δούμε και τον, οικοδομικό, τον κατασκευαστικό τομέα να δούμε δηλαδή κατά πόσο ε, οι ενώσεις εργαζομένων και εργοδοτών είναι υπέρ ανοιχτού καταλόγου. Για το 12 πρέπει να πω ότι θα είναι το δυσκολότερο στην ΙΜΚΟ. Δεν συμφωνούμε για την εξολοκλήρου ευθύνη και την, την αποκοινού ευθύνη. Ε, έχουμε πολλά ακόμη να συζητήσουμε, αλλά κάτι που είπα και σήμερα το πρωί, ο κατακαιρματισμός, ο κατακαιρματισμός υπάρχει ήδη. Ίσως θα έπρεπε να σκεφτούμε την ίδρυση μιας ευρωπαϊκής από κοινού και εξολοκλήρου ευθύνης, αντί να έχουμε 15-20 διαφορετικές τέτοιες ευθύνες. Επίσης, για τα θέματα της διαφάνειας, της ε, πληροφόρησης, καλύτερης συνεργασίας... Ε, και της ε, εξέβρεσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που παραγνωρίζονται πάρα πολύ στο πλαίσιο του σημερινού ανταγωνισμού. Ευχαριστώ. Ρέγνερ και μετά Μπένιον. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Είμαι η συγκητρία της εκνομοδότησης από την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. Προχθές στη συνάντηση των συντονιστών ανακοινώθηκε ε, προχθές μόλις στη συνάντηση των συντονιστών το συζητήσαμε, δεν μπορώ λοιπόν να σας ανακοινώσω κάποια, ε, κάποιες ε, αποφάσεις. Το χρονοδιάγραμμα μας φαίνεται κάπως μικρό, κάπως σύντομο, πρέπει να εργαστούμε πάρα πολύ γρήγορα και ελπίζω να καταφέρουμε να προλάβουμε την ψηφοφορία του Ιανουαρίου και να εμπλουτίσουμε την ε, γνωμοδότηση με τις δικές μας ε, απόψεις. Μας αναφέρατε ότι ασχολείστε με έναν σχετικά στενό τομέα των νομικών ε, απόψεων και φυσικά εμείς θεωρούμε ως νομική επιτροπή ότι το ζήτημα της ευθύνης είναι ιδιαίτερα σημαντικό Τώρα, όσον αφορά την ε, παρουσίαση που μας κάνατε, εγώ καταλαβαίνω το δίκαιο ως εξής. Εδώ μας απασχολεί βέβαια ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι όμως κάτι το οποίο δεν ολοκληρώνεται ποτέ, δεν τελειώνει, πάντα εξελίσσεται και ιδιαίτερα στους τομείς της συνεργασίας, της διοικητικής συνεργασίας, της διασυνοριακής Διοικητική συνεργασία, πρέπει να προσέξουμε ε, να εφαρμοστούν μέτρα τα οποία θα τηρούν το δίκαιο, το ισχύον δίκαιο. Δεν θα αρχίσω να σας τα αναφέρω τώρα από το μηδέν. Σίγουρα θα ξέρετε όλες τις λυπηρές ε, ιστορίες που μας οδηγούν στο να επιστρέφουμε και να έχουμε να αντιμετωπίσουμε δυσάρεστες ε, Ερωτήσω, όπω για παράδειγμα είναι ποια είναι η στάση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τι κάνει το, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τίποτα. Τι κάνει, τι γίνεται με το κοινωνικό dumping, πώς ερμηνεύεται εδώ το κοινωνικό δίκαιο. Χρειάζονται μέτρα που θα φροντίζουν να τηρείται το δίκαιο στα, σε όλα τα κράτη-μέλη. Και τόσοι πολλοί ομιλητές πριν από μένα ανέφεραν ότι είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη και δεν είναι κάτι μεμονωμένο. Υπάρχει ένα ολόκληρο σύστημα και ακριβώ για το λόγο αυτό, ακριβώ για αυτό το background, θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό ε, το ότι έχουμε την εσωτερική αγορά, αλλά επίση είναι εξίσου σημαντικό όλοι μα να δείχνουμε τον ε, δέοντα σεβασμό στην εσωτερική αγορά έτσι ώστε όλοι να μπορέσουμε να ωφεληθούμε από αυτό. Γι' αυτό θα ήθελα να πω στην εισηγήτρια να μην έχει μόνο υπόψη την, την παροχή υπηρεσιών και τις αποσπάσεις, αλλά το γενικότερο πλαίσιο της εργασία... του εργασιακού καθεστώτος που πάσχει από dumping μισθολογικό. Ε, και μετά ο κ. Κλωσόφσκι. Θα είμαι σύντομο ε, γιατί συμφωνώ με τα περισσότερα από αυτά που είπε η εισηγήτρια για την έκθεση, στην έκθεσή της. Για τον κατάλογο εγώ θα προτιμούσα έναν κλειστό κατάλογο, όμως ε, νομίζω ότι δεν χρειάζεται υποχρεωτικά να είναι ο κατάλογος που έχουμε αυτή τη στιγμή. Μπορούμε να το συζητήσουμε αυτό. Ένας από τους τομείς ε, που δεν, με βρίσκει σύμφωνο είναι ο λευκός κατάλογος ε, έμπιστων εταιριών, ε, αξιόπιστων μάλλον, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι ένα προφανές εμπόδιο για νεοεισερχόμενους και θα προτιμούσα να μην ακολουθήσουμε αυτήν την οδό. Το θέμα τώρα της από και εξολοκλήρου ευθύνης το έχω ξαναθήξει σε προηγούμενες συνεδριάσεις και θα προτιμούσα να ακολουθήσω τη διαγραφή. Υπάρχουν τροπολογίες βέβαια στην ΙΜΚΟ που την επιτρέπουν αυτή την ευθύνη που θέλουν να χρησιμοποιήσουν αυτό το σύστημα, κάτι το οποίο είναι, πιστεύω ότι είναι ένας πολύ καλύτερος τρόπος καλό θα ήταν χώρες που δεν έχουν τέτοιου είδους ευθύνη, τέτοιου είδους σύστημα δηλαδή, να, τις, να μην τις υποχρεώσουμε να αποκτήσουν ένα τέτοιο σύστημα θα ήταν καλύτερα, πολύ καλύτερα, να ενισχύσουμε τη συνεργασία μεταξύ του αποσπάζοντος κράτους μέλους, προέλευσης τέλος πάντων και του κράτους υποδοχής, ένα σύστημα ελέγχου όπως είπε και ο κύριος Μαν και να εξασφαλίσουμε ε, ότι ο έλεγχος και η συνεργασία είναι τέτοια ώστε ε, να υπάρχει δίωξη ε, μέσω του νομικού συστήματος αν υπάρχουν προβλήματα και όχι να ιδρύσουμε ένα σύστημα βάσει του οποίου ε, κάποιος πληρώνει την ύφη αν δεν μπορεί να πιάσει αυτόν που έχει κάνει μία παρατυπία. Ε, νομίζω ότι αυτό είναι πολύ καλύτερο. Αν εγώ είμαι ένας επιχειρηματίας που είμαι κατά κάποιο τρόπο, ε, μπορεί να διαλέξω έναν μειοδότη από τη δική μου τη χώρα, επειδή εκεί δεν ισχύει αυτό το σύστημα της από και αξιολοκλήρου ευθύνης, αντί να διαλέξω κάποιον άλλον ε, από μια άλλη χώρα. Κάτι το οποίο νομίζω ότι κάνει πολύ μεγάλη διαφορά αν σημαίνει κάποιο κίνδυνο, ότι θα εκτεθώ δηλαδή σε κάποιο κίνδυνο. Πολλέ χώρε δηλαδή μπορεί να προτιμήσουν το δικό του ε, τον πάροχο αντί τον ξένο. Και δεν νομίζω ότι αυτό είναι καλό για τον ανταγωνισμό. καλύτερα συνεργασία μέσω του νομικού συστήματος για την απόσπαση και για τις χώρες υποδοχής. Νομίζω ότι είναι καλύτερο να διώκονται ε, όσοι κάνουν παρατυπίες ε, από το σύστημα που προτείνεται εδώ. Ο κύριος Κλωσόφσκι και μετά η κυρία Μάκιντάιρ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ίσως αυτό να είναι ε, και η μοίρα όλων των ε, ε, τελευταίων ομιλητών, γιατί ό,τι ήθελα να πω τα είπαν οι άλλοι συνάδελφοι, άρα δεν χρειάζεται να τα επαναλάβω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που είπατε. Η κυρία Μάκιντάιρ. Ευχαριστώ ε, κύριε Πρόεδρε. Chairman στα αγγλικά. Όχι, είμαι chairwoman, λέει η Πρόεδρος. Εξ ονόματος ε, του ECR θα ήθελα ε, να ευχαριστήσω την εισηγήτρια και να συμφωνήσω με τις αρχές τις οποίες έχει καθορίσει στην έκθεσή της. Δεν μιλάμε μονάχα για την δυνατότητα μετακίνησης των εργαζομένων ή κυκλοφορίας των εργαζομένων και την απόσπασή τους. Μιλάμε για την δυνατότητα ε, ελεύθερης παροχής ε, ε, υπηρεσιών. Βεβαίως δεν έχει οργανωθεί η εσωτερική αγορά όσον αφορά τις υπηρεσίες. Προσπαθούμε να το κάνουμε όσον αφορά το άρθρο 5. Συμφωνώ με αυτά που είπε ε, που αναφέρεται στο σημείο αυτό και χαίρομαι που τα έχω στα αγγλικά. Η διαγραφή τώρα του άρθρου 12 θα μπορούσα να συμφωνήσω με αυτό. Ε, πιστεύουμε ότι ένα τέτοιο άρθρο μπορεί να αποτελέσει πρόσκομα ε, για την ελεύθερη κυκλοφορία ε, και τον ανταγωνισμό. Πιστεύω ότι πρέπει να κλείσει το μικρόφωνο της Προέδρου παρακαλούμε, δεν ακούμε καλά. Ευχαριστούμε. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να ε, ε, προστατεύσουμε αυτούς ε, οι οποίοι δεν προστατεύονται από τις εταιρείες τους ή αυτές τις εταιρείες που είναι εταιρείες φραγίδες που δεν υπάρχουν πραγματικά. Έχουν μόνο μια ταχυδρομική θηρίδα. Ε, γιατί διαφορετικά ε, βεβαίως ε, εδώ θα έχουμε και μη προστασία των εργαζομένων και πρόσκομα στην, στον ελεύθερο ανταγωνισμό. Θα, ακόμα δεν έχουμε καθορίσει θέση όσον αφορά τις διοικητικές ποινές και την εφαρμογή των αποφάσεων, αλλά θα προετοιμάσουμε οπωσδήποτε τροπολογίες και ε, θα συνεχίσουμε την τόσο καλή συνεργασία που είχαμε μέχρι τώρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ ε, κυρία Μακιντάρ. Ζητώ συγγνώμη γιατί έκανα σχόλια εντός ε, μικροφώνου, <laughs> ενώ θα έπρεπε να είναι εκτός μικροφώνου, εν πάση περιπτώσει. Ο Αλεξάνδρος Σάρκας. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ξεκινούμε τώρα μία συζήτηση η οποία είναι ε, η οποία σίγουρα δεν θα είναι απλή. Το μαντέψαμε ήδη από τώρα, το είπε και η ίδια η συγγήτρια. Κοιτάξτε, εγώ πρέπει να σας πω σαν σοσιαλιστής ότι εμείς έχουμε συζητήσει επανειλημμένα το θέμα αυτό. Θέλω δύο κριτήρια να μου δώσετε τα οποία θα επιτρέψουν την προσέγγιση των θέσεων μας, αλλά θα πρέπει να αλλάξει η ε, προοπτική βάσει της οποίας έχετε αντιμετωπίσει το ζήτημα αυτό για μας. Ε, θα πρέπει να γίνουν σεβαστοί οι αρχές προστασίας των εργαζομένων. Δεν θέλουμε λιγότερους ελέγχους, δεν θέλουμε να ε, καταστεί δυνατή η ελεύθερη κυκλοφορία των ε, εργαζομένων παρά μόνο εάν καλύπτονται κάποιες ελάχιστες κοινέ ε, προδιαγραφές. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι να υπάρχουν τέτοιοι κανόνες βάσει των οποίων θα αποφεύγονται οι καταχρηστικές διαδικασίες. Κοιτάξτε, η οδηγία έχει νομικές ε, ατέλειες ε, και έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις που αναγκαστήκαμε να φτάσουμε στο δικαστήριο και να χρησιμοποιήσουμε ε, την νομολογία του δικαστηρίου. Έχουμε διαπιστώσει ότι βεβαίως έχουμε και τις εθνικές νομοθεσίες μας οι οποίες μπορεί να ε, ε, διαφέρουν. Βλέπουμε πώς έχει η κατάσταση. Δεν θέλουμε να γίνει ακόμα πιο ευέλικτη η αγορά και δεν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε ε, άρθρα τα οποία δεν έχουν γραφτεί σωστά έτσι ώστε να επιτρέψουμε να εξασθενήσει ακόμα περισσότερο ο σωστός ανταγωνισμός. Από την άλλη μεριά δεν θέλουμε ούτε ρατσιστές να γίνουμε, ούτε ξενόφοβοι, ούτε τίποτα. Θέλουμε κανονισμούς, θέλουμε αρχές, θέλουμε πρόνοια στην οδηγία αυτή, η οποία, οι οποίες να μπορούν να ε, αποσαφηνίσουν την κατάσταση. Αυτή η οδηγία για την απόσπαση των εργαζομένων δεν είναι καλή. Δεν την έχουν γράψει σωστά δεν επιτρέπει ούτε να, να ερμηνεύονται οι αρχές σωστά, ούτε και ε, να αποφεύγονται οι καταχρήσεις. Δεν είναι νέα οδηγία, τη γνωρίζουμε. Θέλουμε τώρα να την επικυροποιήσουμε και να την επιβάλλουμε σωστά. μια απλή οδηγία της Κομισιόν ε, η οποία να ε, προβλέπει την εφαρμογή της οδηγίας, όχι δεν μας αρκεί δεν ναι, μας αρκεί. Θέλουμε ε, τρόπους ελέγχου που να επιτρέπουν ε, τον, τον σωστό έλεγχο. Δεν θέλουμε περαιτέρω ε, αποδυνάμωση των εργαλείων. Επίσης δεν θέλουμε εθελούσιους κανόνες, δεν θέλουμε κανόνες που θα έγκυται στην διακριτική ευχέρεια των κρατών, θέλουμε σωστούς ελέγχους, αποτελεσματικούς ελέγχους. Έχουμε μία σειρά ανθρώπων ε, που δεν ε, ε, ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους. Εμείς δεν θέλουμε να δουλέψουμε κατά των επιχειρήσεων. Εμείς θέλουμε να είμαστε κατά των επιχειρήσεων που τα διαταράσουν την εργασιακή ειρήνη. Είμαστε κατά των επιχειρήσεων οι οποίες διαπράττουν αδικίες και σφάλματα. Είμαστε κατά των επιχειρήσεων οι οποίες προσπαθούν να περιγράψουν το σύστημα σύστημα και οι οποίες προσπαθούν να επωφεληθούν από τα κενά που αφήνουν ε, τα κείμενα. Θέλουμε οδηγία που πραγματικά θα προστατεύει και τους εργαζόμενους και, τους, και τις επιχειρήσεις με την προϋπόθεση ότι θα είναι σωστές και αξιοπρεπείς επιχειρήσεις. Είναι πάρα πολύ δύσκολο πιστεύω να επιτύχουμε σε συμφωνία, ε, να επιτύχουμε συμφωνία, να φτάσουμε σε συμφωνία εάν ε, δεν αλλάξει η, ε, η συγγήτρια την προοπτική με την οποία βλέπει τα πράγματα. Θέλουμε προστασία των εργαζομένων, θέλουμε να τελειώσουμε με αυτές τις πειρατικές πρακτικές. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Μαδεσσαρτιέ, ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την Τανούτα για την εργασία την οποία έχει κάνει. Διαβλέπω την πρόθεσή της να προστατέψει τους εργαζόμενους, χωρίς όμως, Αλεχάνδρο, να καταστραφεί η απασχόληση, γιατί, Αλεχάνδρο, η απασχόληση είναι οι επιχειρήσεις που προωθούν την απασχόληση. Υπάρχει ένα σημείο το οποίο μου φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι η έννοια του ελέγχου. Πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε και κλειστούς καταλόγους κριτηρίων που θα μας δίνουν την δυνατότητα να ε, υπάρχει μια συνεκτική αντιμετώπιση των χωρών, να, να ε, κουμπώνει μια χώρα με την άλλη σε επίπεδο των 27. Εγώ ε, είμαι εξαιρετικά διστακτική ε, στο ενδεχόμενο να δώσουμε τη δυνατότητα στα κράτη να προσθέσουν ε, κριτήρια, γιατί είναι βέβαιο ότι με τον τρόπο αυτό θα προσπαθήσουν να αποδυναμώσουν κριτήρια τα οποία υπάρχουν ήδη ε, στον κατάλογο. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει οι κατάλογοι των κριτηρίων να είναι κλειστές και μόνο βάσει αυτών των καταλόγων ε, να γίνεται ο έλεγχος. κάθε ελεγκτής θα σας πει ότι εάν δεν υπάρχουν συγκεκριμένα και Σαφώ καθορισμένα κριτήρια δεν μπορεί να υπάρχει σωστός έλεγχος. Το είπα και το πρωί για την έκθεση του Στέφεν Χιούξ. Εάν θέλουμε να έχουμε μία σωστή και κοινή κοινωνική πολιτική σε ευρωπαϊκό ενωσιακό επίπεδο θα πρέπει να αρχίσουμε να σφίγγουμε λίγο τις βίδες. Αυτό πρέπει να αρχίσουμε να κάνουμε, να σφίγγουμε τι βίδες. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε εδώ τον παλιό μα συνάδελφο συζητητή της Επιτροπής των Περιφερειών. τον συνάδελφο Χάτζινσον. Δεν μας ενδιαφέρει εδώ να συζητάμε περί ανέμων και υδάτων για μια ε, οδηγία και θέλουμε να την ε, αλλάξουμε, να την τροποποιήσουμε. Θέλουμε να προβλέψουμε τις επιπτώσεις και να αποφύγουμε τις κακές επιπτώσεις. Εδώ, και ζυγίζω πολύ καλά τα λόγια μου, Νομίζω ότι όταν μιλάμε για αυτά τα ζητήματα ε, είναι σαν να μιλάμε για την Ευρωζώνη και σαν να μιλάμε ε, και για τις μελέτες αντικτύπου στην ε, Ευρωζώνη. Ελάτε λίγο στη χώρα μου δέστε τι γίνεται κυρίως στα εργοτάξια, είναι πόλεμος, γίνεται πόλεμος. Οι Γάλλοι εργαζόμενοι δεν είναι ότι στρέφονται κατά του των Πολωνών ε, υδραυλικών. Απλώς δεν μπορούν να ανεχτούν οι Πολωνέζοι, οι Ιδραυλικοί, οι Σλοβάκοι, οι Γερμανοί οποιοδήποτε να έρχονται να εργάζονται στη Γαλλία χωρίς να σέβονται τους κανόνες ασφάλειας, υγιεινής, χρόνου εργασίας, κοινωνικής προστασίας, ε, μισθού κτλ. της χώρας υποδοχής. Εκεί είναι η συζήτηση. η συζήτηση που είχαμε όταν συζητούσαμε την οδηγία για τις υπηρεσίες και ξαναρχίζει η συζήτηση αυτή σήμερα. Και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια κατάσταση ε, εντονότητα της κοινωνικής έντασης, μεγάλης κοινωνικής έντασης. Επομένως δεν είναι τώρα λόγος για να κάνουμε συζήτηση για τα α, β, γ δικαιώματα ή υποδικαιώματα κτλ. Εδώ έχουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση στην οποία και τα αγαθά και οι άνθρωποι μπορούν να κυκλοφορούν ε, ελεύθερα. Υπάρχει ίσω μια νομική βάση την οποία έχετε καταδείξει, αλλά εμεί σαν πολιτικοί υπεύθυνοι δεν είναι δυνατόν να δούμε την οδηγία αυτή ξέχωρα από την κοινωνική προστασία των εργαζομένων, γιατί διαφορετικά τελικά οι ίδιοι εργαζόμενοι θα στραφούν μαζικά κατά τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Λυπάμαι που λέω τόσο μεγάλα και βαρύγδουπα λόγια, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι το διακύβευμα εδώ. Αυτό συζητούμε και δεν είναι καθόλου μικρό αυτό που έχουμε απέναντί μα. Είναι τεράστιο το εύρο του θέματος που μας απασχολεί και επομένως ορισμένες προτάσεις σα, τι να σα πω, με, με, με, με εκπλήσουν. Ε, ξέρω ότι ήθιστε να λέμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον εισηγητή για τη δουλειά που έκανε. Εγώ δεν θα το πω, δεν θα το πω. Ε, ε, έχουμε τώρα αυτό το άρθρο 12 το οποίο διαγράφεται και το οποίο αφορά τις υπεργολαβίες, αφορά την ευθύνη ε, από κοινού και εξ ολοκλήρου. Μα δεν είναι δυνατόν αυτό να, με μία μονοκοντιλιά να το διαγράψουμε προτείνετε μας, εν πάση περιπτώσει, έστω κάποια εναλλακτική διατύπωση και δεν στρέφομαι λέγοντας αυτό κατά των ε, εργαζομένων. Πιστέψτε με σας παρακαλώ. Το λέω εξ ονόματος όλων των εργαζομένων και για την προστασία όλων των εργαζομένων. Θα πρέπει να ξεφύγουμε από την από το αδιέξοδο στο οποίο έχουμε οδηγηθεί με αυτήν την οδηγία για, τους, ε, για την απόσπαση των εργαζομένων. Και δεν μιλάμε μονάχα για τους μισθωτούς, μιλάμε για όλους τους εργαζόμενους. Επομένως θα καθίσουμε εδώ όσο χρειάζεται για να συζητήσουμε ενδελεχώς το ζήτημα, γιατί ε, έχουμε τις εκλογές το 2014 και με τι μούτρα θα δούμε τους ε, ψηφοφόρους μας το 2014 πριν τις εκλογές. Δεν θα μπορούμε να τους κοιτάξουμε στα μάτια. Λοιπόν, καταλαβαίνω πώς σκέφτεται η Ντανούτα, αλλά εγώ ε, δεν μπορώ να ε, ε, μην συζητάω, να μην λέω αυτά που σκέφτομαι. Όσον αφορά τώρα την επιθεώρηση εργασίας, τους ελέγχους, και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Όταν θα καθορίσουμε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο, θα, α, γιατί να, να σας πω, εδώ πέρα διαρριγνούμε τα ημάτια μας και λέμε ότι θα πρέπει να υπάρχει εποπτεία των κεφαλαίων θα πρέπει να υπάρχει εποπτεία των διακινουμένων κεφαλαίων κτλ. κτλ. Εδώ δεν πρέπει να υπάρχει έλεγχος, δεν πρέπει να υπάρχει εποπτεία. Ευχαριστώ πολύ κυρία Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Μετά από αυτά τα που είπατε δεν νομίζω ότι υπάρχει περιθώριο για να πω και εγώ πολλά. Όπως είπατε ε, προηγουμένως είμαι εισηγητής για την ε, εξέταση της προτάσεως οδηγίας αυτής στην Επιτροπή των Περιφερειών. Ε, αύριο στην Ολομέλεια της Επιτροπής των Περιφερειών που θα λάβει χώρα εδώ στα κτίρια του Κοινοβουλίου θα εγκριθεί το σχέδιο γνωμοδότησης το οποίο έχει ήδη μελετηθεί η Επιτροπή των Περιφερειών στόχο έχει να ε, ε, προσπαθήσει να απαντήσει σε τέσσερις κύριους στόχους, κύρια κεντρικά μελήματα, τα οποία θα σας ε, αναφέρω εν συντομία. Πρώτον, ε, να αξιολογήσουμε ε, τον ρόλο των ε, κοινωνικών εταίρων όσον αφορά την απόσπαση των εργαζομένων, γιατί αυτό λείπει. Δεύτερον, να αποφύγουμε πάση θυσία να αμφισβητήσουμε ή να θέσουμε ένα αμφιβόλο το πνεύμα της οδηγίας του 71. Τρίτον, να προστατέψουμε τα δικαιώματα των αποσπασμένων εργαζομένων και τέταρτον, να διασφαλίσουμε την ενσωμάτωση της οδηγίας όταν θα έχει εγκριθεί. Ε, όσον αφορά το πρώτο θέμα του κοινωνικού εταίρους, ε, θέλουμε τροποποίηση τη νομική βάση. Η νομική βάση η οποία χρησιμοποιείται στην πρόταση της ε, Κομισιόν αφορά την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών. Εμεί επιθυμούμε η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων να αναφερθεί και να ληφθεί ως νομική βάση τη εν λόγω οδηγία. Η πρόταση οδηγίας ενδιαφέρει άμεσα και την εφαρμογή των κανόνων εργασία ε, Συλλογική διαπραγμάτευση διαπραγμάτευσης, κατώτατη αμοιβή και επομένως ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο τουλάχιστον θα πρέπει να υπάρχει διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους. Ε, πολλό δε μάλλον που αναφέρεται ρητά στην οδηγία ο ρόλος που μπορούν οι κοινωνικοί εταίροι να παίξουν όσον αφορά το σεβασμό των κανόνων. Το δεύτερο σημείο για, όσον αφορά την σωστή επιβολή της οδηγίας 96 του 71. Ε, στην παρούσα πρόταση της ε, Επιτροπής γίνεται μια προσπάθεια ε, να απομακρυνθεί από το πνεύμα της Οδηγίας 9671. Υπάρχουν κάποιες υποχρεώσεις τις οποίες η Οδηγία 9671 ασκούσε επί τρίτων χωρών και όχι μονάχα επί των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να επανέλθουμε σε αυτή τη διατύπωση έτσι ώστε να αποφύγουμε οποιαδήποτε μορφή κοινωνικού ντάμπινγκ από τρίτες χώρες γιατί ξέρουμε ότι αυτό υπάρχει. Και επίσης να ληφθούν υπόψη διατάξεις οι οποίες αφορούν ε, το άρθρο 8 της Ρώμη 1 ε, που αναφέρονται και στην ε, οδηγία του 96, την οδηγία 9671 καθώς επίσης και στην οδηγία για τις υπηρεσίες που τότε που ήμουν ακόμα στο Κοινοβούλιο είχα την τιμή να ασχοληθώ με την οδηγία αυτή. Αυτά είναι τεχνικά στοιχεία ενδεχομένως, τα οποία όμως τελικά καταλήγουν σε ιδιαίτερα σημαντικά κοινωνικά διακυβέρματα. Τρίτον, ενίσχυση του ελέγχου των αποσπαζόμενων εργαζομένων. Ε, ε, εμείς εδώ προτείνουμε ένα περιορισμό όσον αφορά την κάθετη υπεργολαβία ε, εν είδη καταράκτη, δηλαδή της διαρκής συνεχής Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι από ένα σημείο και πέρα υπεργολαβία βία στην υπεργολαβία. Είναι αδύνατον να ελέγξουμε την κατάσταση. Έχουμε και εδώ στο Βέλγιο, στην Μάρσο Αμφλανέλ, ε, έχουμε καμιά πενταριά εργαζόμενους βούλγαρους που δουλεύουν ε, σε, αυτήν την, ε, σε αυτό το κατασκευαστικό εργοτάξιο που δεν ξέρω κι εγώ πόσους μήνες έχουν μείνει απλήρωτοι γιατί δεν μπορούμε να βρούμε ποιος είναι ο αρχικός εργολάβος. Από υπεργολάβο σε υπεργολάβο είναι αδύνατο να ανεβούμε στην αλυσίδα των υπεργολάβων και τελικά καταλαβαίνουμε ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ περίπλοκη. Επίσης οι εκπρόσωποι των εργαζομένων εργαζομένων, κυρίως δε τα μέλη ε, της, ε, των Ευρωπαϊκών ε, Επιχειρησιακών Συμβουλίων θα πρέπει να έχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Τέλος, πιστεύουμε ότι θα πρέπει, για το τέταρτο σημείο τώρα, θα πρέπει να υπάρχει στην οδηγία πρόβλεψη η οποία θα αναφέρεται στην εξολοκλήρου και από κοινού ευθύνη όσον αφορά την υπεργολαβία και αυτό θα πρέπει να είναι δέσμευση ότι θα αναφέρεται ρητά και στην ενσωμάτωση της οδηγίας στα εθνικά δίκαια των κρατών μελών. Αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά ζητήματα και να μην ξεχνούμε ότι πίσω από αυτή την οδηγία, πίσω από αυτά που συζητάμε εμείς σήμερα, κρύβονται εκατομμύρια άνθρωποι, εκατομμύρια εργαζόμενοι. Και ο Γάλλος ε, Υπουργός ε, ε, Απασχόλησης είπε πρόσφατα ότι ε, στην ε, Γαλλία έχει δεκαπλασιαστεί από το 2006 ο αριθμός των αποσπασμένων εργαζομένων. Στην, ε, στο Βέλγιο αυτή τη στιγμή ισχύει περίπου το ίδιο. Έχουμε καμιά 300.000 εργαζόμενους και δεν είναι δυνατόν να επιτρέψουμε να έρχονται εδώ άνθρωποι, Πορτογάλοι ή οποιασδήποτε άλλη εθνικότητα που θα δουλεύουν στο Βέλγιο και δεν θα έχουν τι ίδιε κοινωνικέ παροχέ και λοιπέ παροχέ με του Βέλγου εργαζόμενου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μας ενημερώσατε για τη δική σας γνωμοδότηση που θα ψηφιστεί αύριο ε, στην Επιτροπή Περιφερειών. Δέκα λεπτά μας μένουν για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για την εισηγήτρια. Δεν είναι επαρκής ο χρόνος, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να ολοκληρώσουμε σε δέκα λεπτά, γιατί διαφορετικά αύριο το πρωί ε, θα πρέπει να αρχίσουμε με αυτό το θέμα ή την επόμενη φορά. Ο κύριος Σίλβα Πέντε λεπτά εσείς λοιπόν και πέντε λεπτά η συγγήτρια. Ευχαριστώ πολύ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε ήδη την ευκαιρία να παρουσιάσει την πρόταση αυτή στην προηγούμενη ακρόαση, οπότε σήμερα δεν θα μπω σε λεπτομέρειες και θα είμαι σύντομος. Θα ήθελα να κάνω μερικά σύντομα σχόλια. Καταρχά, να σα υπενθυμίσω ότι με την πρόταση αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποσκοπεί στο να ενδυναμώσει την κοινωνική διάσταση τη ενιαία αγορά και να επαναφέρει την εμπιστοσύνη ανάμεσα στους ενδιαφερομένους με, δίδοντας περισσότερη διαφάνεια και σαφήνεια. Έπειτα θέλουμε να αποτρέψουμε την κατάχρηση των κανόνων και να θεσπίσουμε μία δίκαιη κατάσταση για όλους τους ενδιαφερομένους. Επιπλέον να διασφαλίσουμε ότι οι εργαζόμενοι θα πληρώνονται. Και εδώ θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι στόχος μας και σκοπός μας δεν είναι να επανέλθουμε στην ε, προηγούμενη οδηγία, διότι κάποια από τα δικαιώματα που έχουν δοθεί στους αποσπασμένους εργαζόμενους δεν έχουν εφαρμοστεί στην πράξη. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω πως δεν είναι καλή ιδέα να προσθέσουμε περισσότερα δικαιώματα στην οδηγία, αφού ξέρουμε ότι τα δικαιώματα που ήδη προβλέπονται δεν γίνονται σεβαστά. Με αυτή την εφαρμοστική οδηγία αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να δώσουμε περισσότερα μέσα ελέγχου και περισσότερη σαφήνεια. Δεν δίνουμε προτεραιότητα στις αρχές της χώρας προέλευσης. Το αντίθετο όμως θεσπίζουμε με ξεκάθαρα τρόπο τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της χώρας ε, υποδοχής και της χώρας προέλευσης. Και προτείνουμε ένα λεπτομερές σύστημα συντονισμού ανάμεσα στις αρχές πολύ περισσότερο λεπτομερές από ό,τι προβλέπεται στην ισχύουσα οδηγία 96 71 όπου δεν υπάρχουν πρακτικοί κανόνες. Αυτό λοιπόν προσπαθούμε να κάνουμε, να βελτιώσουμε το σύστημα συνεργασίας. Τώρα, έχουμε παρατηρήσει τις συζητήσεις στο Συμβούλιο, έχει επιτευχθεί κάποια πρόοδος είναι η αλήθεια και φυσικά ε, παρακολουθούμε τις εξελίξεις αυτήν εδώ την Επιτροπή θα ήθελα όμως να αφήσω το εξή μήνυμα. Πρόθεσή μας είναι να δημιουργηθεί μια, ένα σύνολο ισορροπημένων κανόνων. Μια ισορροπία ανάμεσα στα δικαιώματα των εργαζομένων, ιδιαίτερα των αποσπασμένων και την προστασία των, ε, επιχει... των των επιχειρήσεων να ε, ε, κάνουν διασυνοριακές εργασίες. Και αυτή η ισορροπία έχουμε παρατηρήσει πως έχει ορισμένα εμπόδια και, και στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο θεωρώ πως πρέπει να παραμείνουμε, να, παρα, να ε, παραμείνουμε εστιασμένοι στην επίτευξη της ισορροπίας αυτής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ που ήσασταν σύντομος. Τελειώνουμε με την παρέμβαση της κυρίας Γιαζ, Γιαζουβιέτσκα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να επαναλάβω μετά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι το περιθώριό μας είναι περιορισμένο γιατί δεν μπορούμε να πάμε πέρα από την οδηγία 96 και πρέπει να έχουμε εξισορροπημένους κανόνες. Είμαι υπέρ της αποσαφήνισης όλων αυτών των διατάξεων που εξασφαλίζουν την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων και να αποκλείουμε βεβαίως τους ε, ε, τίμιους εργαζομένους όταν έχουμε έναν εργοδότη που βρίσκεται στην αγορά, στην ε, χώρα υποδοχής και έχει έναν αριθμό, ε, έναν ε, αριθμό προϋποθέσεων τις οποίες πρέπει να πληρεί, χαρτιά να συμπληρώσει. Νομίζω ότι πρέπει να, ισχύει, να ισχύουν οι ίδιοι, οι κανόνες ε, για τις επιχειρήσεις που αποσπούν τους εργαζομένους τους. Γι' αυτό εγώ θα ήθελα να εισαχθούν αυτά τα στοιχεία που εξασφαλίζουν την ασφάλεια των εργαζομένων, αλλά είμαι υπέρ της, του κλειστού καταλόγου. Εγώ είμαι υπέρ της εφαρμογής των εθνικών πρακτικών, μια και μιλάμε στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς ε, και μάλιστα τη συστήνω όταν πρόκειται για ελέγχους. Είμαι της απόψεως ότι θα έπρεπε να μιλούμε για τη διαφάνεια των πρακτικών αυτών και την, ε, τις πληροφορίες ώστε να εξασφαλίζονται ε, τα δικαιώματα των εργαζομένων και ο εργοδότης να γνωρίζει πλήρως τις υποχρεώσεις του. Ποτέ δεν είπα εγώ να αποφύγουμε τους ελέγχους ή να, αυξήσουμε τον αριθμό των ελέγχων. Εγώ νομίζω ότι ε, ο έλεγχος είναι ένα βασικό μέτρο που θα έπρεπε να είναι ανάλογο με... να υπάρχει δηλαδή μια αναλογικότητα σε σχέση με τους εργαζομένους τους υπόλοιπους στη χώρα υποδοχής. Το άρθρο 12 δεν αλλάζει το πώς έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Σε 8 κράτη-μέλη υπάρχει το σύστημα της αποκοινού και ισολόκληρων ευθύνη και η διαγραφή του άρθρου 19 δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει εφαρμογή αυτού του συστήματος. Εγώ λέω να το διαγράψουμε γιατί δεν θέλω να καταλήξουμε σε μια κατάσταση στην οποία θα γινόταν η εισαγωγή αυτού του συστήματος ευθύνης μόνο ε, για τους εργοδότες που αποσπούν τους εργαζομένους τους. Θέλω να αποφευχθεί αυτή η κατάσταση βάσει της οποίας μπορεί κάποιος να διαλέξει τον ε, υπεργολάβο του και να διαλέξει μάλιστα εκείνους όπου δεν υπάρχουν δυσανάλογοι κανόνες. Θα ήθελα να τονίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, τη διαγραφή του άρθρου 10 και να λέει ότι αυτό, να αναφέρεται μάλιστα ότι αυτό διατηρεί την κατάσταση όπως έχει αυτή τη στιγμή στα κρατη Για την εισαγωγή της χώρας ε, υποδοχής και του ορισμού της. Πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η πρόταση και περιμένω σαφή και συγκεκριμένη διατύπωση εκ μέρους σας. Επίσης, αναφερθήκατε στην αποσαφήνιση των σχέσεων μεταξύ των γραφείων ε, ευρέσεως εργασίας. Εμείς προτείναμε διατάξεις οι οποίες ε, σε κάποιο βαθμό θα μπορούσαν να περιορίσουν αυτή, αυτές τις ε, αυτές τις εταιρείες που έχουν απλώς μια ταχυδρομική θηρίδα. Μιλάω για το 1 α Δεν θέλουμε να ιδρύονται τέτοιου είδου εταιρείε. Μία ταχυδρομική θηρίδα είναι πάρα πολύ επικίνδυνο κάτι τέτοιο. Επίσης, κύριε Χιούζα, αναφερθήκατε σε ένα νέο κατάλογο κριτηρίων βάσει του οποίου μπορούμε να, βρούμε, να δούμε κατά πόσο κάποιος είναι αυτοαπασχολούμενος ή όχι σε μια δεδομένη χώρα. Πολύ ενδιαφέρουσα και αυτή η πρόταση. Βεβαίως θα λάβουμε υπόψη τέτοιου είδους τροπολογίες. Η διαγραφή του άρθρου 12 διατηρεί την κατάσταση όσο έχει αυτή τη στιγμή. Νάντια Χίρς. Και εγώ θα ήθελα, και από περιμένω μια σύσταση, μια πρόταση. Πώς θέλετε να συμπληρώσουμε αυτή τη δυνατότητα διαγραφής ε, αυτών των τίμιων εργοζεωμένων ε, και των τίμιων εταιριών. Άρθρο 5 και άρθρο 12 ευχαρίστως να τα συζητήσω περαιτέρω μαζί σας. Για τις καλές πρακτικές. Τις έχουμε συζητήσει πολλές φορές για τις εμπειρίες σας. Ε, προσπαθούμε να τις συμπεριλάβουμε. Αναμένω εναγωνίως ε, την πρόταση για νέες προθεσμίες. Στην Πολωνία λέμε ότι δεν πρέπει να βιαζόμαστε, δηλαδή όποιος βιάζεται σκοντάφτει. Χρειαζόμαστε καλές πληροφορίες, καλά δεδομένα μία εταιρεία που απασχολεί χίλια άτομα και αποσπά 200 σε άλλη χώρα και ξαφνικά πρέπει να την κλείσει αυτή η εταιρεία γιατί έχουν κάνει κάποια λάθη. Τι να σας πω, το βρίσκω λίγο απερβολικό. Κυρία Στάινροκ. Με ενδιαφέρει η εμπειρία σας ναι στον ιστότοπο με τις πληροφορίες, γιατί και αυτό είναι ένα, ένας τρόπος ελέγχου ε, για τις εταιρείες. Γιατί αγγλικά, γιατί είναι ευκολότερο να ζητήσει κάποιο από το γιο του ή την κόρη του να μεταφράσουν κάτι από τα αγγλικά. Γι' αυτό εγώ πρότεινα τα αγγλικά. Υπάρχει το πρόβλημα του social dumping. Θα ήθελα να τονίσω ότι οι συνθήκες εργασίας για τους αποσπασμένους, όπως ορίζονται από τα κράτη-μέλη, πρέπει να πληρούνται από τη χώρα υποδοχής. Είναι δικό μας πρόβλημα να μην επιτρέψουμε μέσω των συνθήκων που θα επιτρέψουμε, να μην επιτρέψουμε το social dumping, το κοινωνικό dumping. Συγγνώμη, συγγνώμη πρέπει να σας διακόψω, έχουμε Πρέπει να ολοκληρώσετε, λέει η ε, κυρία Πρόεδρος, ε, γιατί πρέπει να πάμε σε άλλη αίθουσα. Δύο λεπτά, λέει η Πρόεδρος, ένα τελικά της δίνει της ε, κυρίας εισηγήτριας. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Μιλήσατε για τον ιστότοπο, τα μέτρα ελέγχου. Εγώ είμαι απολύτως υπέρ ε, αυστηρών ε, μέτρων ελέγχου. Αλλά ποια είναι αυτά τα μέτρα, πρέπει να τα ξέρουμε. Αλεχάνδρο, θα ήμουν ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος στον κόσμο αν μπορούσαμε να βρούμε έναν τέλειο τρόπο να προστατεύσουμε τους εργαζομένους. Αλλά έχουμε 27 διαφορετικά συστήματα, γιατί έχουμε 27 διαφορετικές χώρες και 27 διαφορετικές εμπειρίες. Προσπαθώ να βρω την καλύτερη λύση. Αν έχεις μια καλύτερη πρόταση, σε παρακαλώ, να μου τη γνωστοποιήσεις. Συγγνώμη. Μπορώ να σα ξαναδώσω το λόγο αύριο, αν θέλετε, λέει η πρόεδρο, στην άλλη μα συνεδρίαση, αλλά πρέπει να σταματήσουμε τώρα. Συγγνώμη που σα διακόπτω, αλλά τι να κάνω, πρέπει να πάμε στην άλλη αίθουσα. Ζητώ συγγνώμη από την ησυχήτρια. Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών 13 Δεκεμβρίου, 12 το μεσημέρι. Έτσι έχει το χρονοδιάγραμμα τουλάχιστον αυτή τη στιγμή. Θα εξετάσουμε τι τροπολογίες στις 23 και 24 Ιανουαρίου. Θα έχουμε συμβιβαστικές τροπολογίες στις 20 Φεβρουαρίου. Εξ, ε, ε, ε, έγκριση στις 21 Φεβρουαρίου. Και θα πάμε στην Ολομέλεια του Μαΐου. Θα ψηφιστεί στην Ολομέλεια του Μαΐου. Πρέπει να πάμε στην κοινή μας συνεδρίαση τώρα. για την παρουσίαση της ετήσιας ε, έκθεσης ανάπτυξης από τους δύο επιτρόπους, Άντορ και Ρεν, στο 4Q1, στην αίθουσα 4Q1. Σας ευχαριστώ πολύ. Τα λέμε εκεί.